Good afternoon, dear ladies and gentlemen. Καλησπέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Να περάσουμε στην απογευματινή μας συνεδρία. Τρεις η ώρα το απόγευμα είναι, 16 Ιουνίου του 2015. Έχουμε την ανάπτυξη βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας κοινών μετάλλων. Ο Έντουαρ Μαρτάν είναι ο συνάδελφος που έχει αναλάβει το θέμα αυτό, η συγκητής μας. Στις 6 Μαΐου μας είχατε παρουσιάσει ένα έγγραφο εργασίας για το θέμα αυτό. Θα κληθούμε σήμερα να συζητήσουμε αυτό το θέμα, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την βιομηχανία μας Χωρίς τα κοινά μέταλλα δεν μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση της οικονομίας μας. Και είμαστε και πολύ εξαρτημένοι από τις εισαγωγές των μετάλλων αυτών, κυρίως από την Κίνα. Και δεν είναι δύσκολη αυτή η κατάσταση για μας. Ο συνάδελφος λοιπόν ε, είναι ο πλέον ειδήμων για το θέμα αυτό ως εισηγητής, οπότε θα ήθελα να του δώσω και το λόγο για να μας πει, να μας κάνει τα σχόλιά του. Ευχαριστώ πολύ Κύριε Πρόεδρε, πριν αρχίσω ε, να, να, κάνω την εισαγωγή για την εξέταση, για την... το σχέδιο έκθεσης που σας έχω υποβάλει, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που με βοήθησαν, με υποστήριξαν ε, για ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτή η βιώσιμη ευρωπαϊκή βιομηχανία κοινών μετάλλων. Να ευχαριστήσω τη Ζαν, τη Μαξί, τον Μαξίμ, τον Φιλίπ, ε, την ομάδα μου που με βοήθησαν πάρα πολύ και που κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να είναι πραγματικά ποιοτική αυτή η έκθεση. Και να μπορέσει να παρουσιάσει όλα τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Τι προσπαθήσαμε να κάνουμε. Ξεκινήσαμε από μια διαπίστωση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Σήμερα η κρίση μας το έχει ε, δείξει αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δώσαμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στη θέση ε, της βιομηχανίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία βασίζεται και στις μεθόδους παραγωγής ε, εκατοντάδες εκατομμύρια τόνων ε, παράγονται κάθε χρόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μιλάμε δηλαδή για παραγωγέ που είναι στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιδέα μα ήταν λοιπόν πώ ακριβώ θα μπορέσουμε να προσανατολίσουμε την ε, ευρωπαϊκή μα πολιτική με τον κίνδυνο τη ε, μείωση των θέσεων εργασία και επίση υπάρχει και το θέμα τη αυτονομίας μας ε, για, από, ε, από ε, ε όπως είναι τα κοινά μέταλλα ε, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη βιομηχανία μας. Πώς λοιπόν μπορούμε να λάβουμε μέτρα ώστε να περάσουμε σε έναν ενάρετο κύκλο από ένα φαύλο κύκλο. Λοιπόν, επί της μορφής να σας πω ότι δεν ε, ε, ήταν προσωπικές οι απόψεις που εκφράστηκαν. Ξεκινήσαμε από μια συγκεκριμένη βάση, από ε, επιτόπου ξεκινήσαμε από τους τοπικούς παράγοντες, ε, επιχειρήσεις, συνδικάτα, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, γιατί ε, το θέμα της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος είναι ένα σημαντικό, μια σημαντική πτυχή. Ξεκινήσαμε λοιπόν από κάτω προς τα πάνω και πρόκειται για μια έκθεση που λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι τοπικοί παράγοντες. Υπάρχει το θέμα του ε, διοξιδίου του άνθρακα. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα να ε, μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτήν την, το επιπλέον κόστος που να μετακυλίεται ε, στους πελάτες, το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας διακυβεύεται. Οπότε αυτό που προτείνουμε είναι το εξής και είναι κάτι το οποίο βρίσκει όλους σύμφωνους, όλους όσους ε, ήρθαμε, όλους, όλους τους ε, συνομιλητές μας. Πρέπει να υπάρχει μια ισότιμη μεταχείριση, να υπάρχει σε διεθνές επίπεδο, ε, στο διεθνή ανταγωνισμό, ένα, μια ισότιμη μεταχείριση, γιατί το βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, πολλές φορές ε, ε, περιορισμοί, υπάρχουν προδιαγραφές που μας δημιουργούν ορισμένες φορές κάποιους περιορισμούς και αυτοί οι περιορισμοί δεν βαρύνουν άλλους παράγοντες, άλλους παίκτες στο διεθνές προσκήνιο όπως είναι οι Κινέζοι για παράδειγμα. Σας υπενθυμίσω ότι ο Wolfgang Έντερ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος Επιτροπής Wall Steel, ανέφερε προχθές ότι αν συνεχίσουμε έτσι ε, η, ε, οι ψυκάμινοι θα εξαφανιστούν ε, στο μέλλον και όχι σε τόσο μακρινό μέλλον. Κάτι λοιπόν, μια τουλάχιστον στρατηγική προσωρινή, ευέλικτη, αν αύριο μπορούμε να βρούμε μια διεθνή συμφωνία και ε, μπορούν όλοι να σέβονται τη διεθνή αυτή συμφωνία. Δεν θα χρειαζόμαστε αυτή την προσαρμογή. Μέχρι τώρα έχουμε κερδίσει το στίχημα της μείωσης ε, ε, του διοξιδίου του άνθρακα, επομένως της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Όλοι οι συνομιλητές μας επέμειναν επίσης στη σημασία του να μπορούμε να έχουμε ε, συμβάσεις ε, ε, μακροπρόθεσμες γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα, για παράδειγμα το κόστος του ηλεκτρισμού είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την προοπτική επενδύσεων των επιχειρήσεων. Σε πολλές χώρες είναι ετήσια αυτά τα συμβόλαια και είναι ένα πρόβλημα για τις επενδύσεις. Αν αύριο είχαμε τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να έχουμε πιο μακροχρόνιες συμβάσεις 10-15 ετών που γίνεται σε άλλα μέρη του κόσμου, οι ίδιοι ε, οι βιομηχανοί μας έλεγαν ότι είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να ευνοήσει τις επενδύσεις. Η εμπορική άμυνα. Όταν υπάρχει ένα σχέδιο anti-dumping, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παίρνει πάρα πολύ χρόνο μέχρι να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις καταγγελίες και ε, τα προϊόντα ε, για τα οποία, τα είναι το αντικείμενο κάθε φορά της εξέτασης μπορεί να εξακολουθούν να διεισδύουν σε ευρωπαϊκές ε, αγορές και να δημιουργούν πρόβλημα στους δικούς μας, στη δική μας βιομηχανία και κάτι ακόμη το οποίο, δεν θα μακρηγορήσω γιατί το διαβάσατε υποθέτω, κάτι ακόμη που μας φαίνεται εξαιρετικά σημαντικό είναι το θέμα της, ε, των αγορών, των κατάλληλων αγορών. Ε, τι έγινε για παράδειγμα στο Τέρνη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αρνήθηκε αυτήν την εξαγορά γιατί θεωρήθηκε ότι ε, το κόμπο θα ήταν σε δεσπόζουσα θέση οπότε πρέπει λοιπόν να ε, ε, ορίσουμε εκ νέου τι θα πει η ε, κατάλληλη αγορά. Κατά τη γνώμη μας αν δεν γίνει αυτό υπάρχει περίπτωση η δική μας βιομηχανία να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με άλλους ανταγωνιστές της όπως στην περίπτωση για παράδειγμα του Τέρνη και την περίπτωση του Οτοκόμπου γιατί υπήρξαν τεράστιες εισαγωγές ε, ανοξίδωτων από την Κίνα και αυτό είχε δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Αυτές λοιπόν ήταν, ε, αυτές οι τέσσερις πυλώνες της εκθεσής μου και είμαι βεβαίως στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε για τα εισαγωγικά σας ε, σχόλια. Να ευχαριστήσω και εγώ τον συνάδελφο Μαρτέν για την έξεση του. Θεωρώ ότι είναι μία έξεση που αποτελεί πολύ μεγάλη ε, στροφή αλλαγή για εμάς εδώ στην Επιτροπή. Περιγράφει ακριβώ την κατάσταση γιατί μιλάμε για μια τεράστια μείωση της παραγωγής στον τομέα του αλουμινίου. Ε, που έχουμε από την πλευρά και από την άλλη την επιβάρηση του περιβάλλοντος. Οπότε οδηγούμε σε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Μέσα από διαφορετικές ε, καταστάσεις οδηγούμαστε στην απώλεια της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως ε, περιέγραψε και ο συνάδελφος Μαρτέν, αυτό έχει να κάνει και με, την, ε, με το διοικητικό φόρτο, ε, κάτι που δυσχεραίνει και τον ανταγωνισμό με άλλα κράτη. Επομένω αυτή η έκθεση θεωρώ ότι αποτελεί μεγάλο σημείο καμπή. Η αξία των ε, βασικών μετάλλων, του αλουμινίου, του χάλιβα κτλ. Οι αξίε του δεν έχουν και πολλές ευκαιρίε. Υπάρχει κίνδυνο σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε μεγάλη εξάρτηση όπως έχουμε σήμερα στον τομέα το πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Πρέπει λοιπόν να αναλογιστούμε την κατάσταση. Κάνουμε λόγο για τις εκπομπές και τον στόχο που πρέπει να, επι... να πετύχουμε. Έχουμε ήδη πετύχει πολλά στον τομέα των εκπομπών. Έχουμε τους κύκλους καινοτομίας, Ε, κύκλους ε, ζωής του αλουμινίου ε, που έχουν σταματήσει ουσιαστικά πριν στο τέλος τους και δεν έχουμε παράλληλα επαρκείς επενδύσεις για εξχρονισμό σε αυτό τον τομέα. Πώς μπορούμε αυτά τα μέτρα, το αλουμίνιο, το χάλιβα και τα πυλά και τα λοιπά να τα παράγουμε χωρίς να επιβαρύνουμε το περιβάλλον. Ένα θέμα μου δημιουργεί ε, ανησυχίες και είναι μια ρύθμιση στον τομέα της διοίκησης είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί στα σύνορα. Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία πλευρά και από την άλλη. Και από την άλλη, τις πιέσεις που μας ασκούνται για τις εκπομπές, ε, να τα συνδυάσουμε και να ε, μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τις εκπομπές χωρίς να έχουμε προβλήματα. Θεωρώ ότι είναι πολύ κέριο λοιπόν αυτό το έγγραφο, αυτή η έκθεση. Με απασχολούν φυσικά τα μέτρα στα σύνορα, αλλά η βιομηχανία, όπως και να έχει, είναι όλο και λιγότερο ανταγωνιστική και γι' αυτό θα ήθελα να εργαστώ περαιτέρω σε αυτή την ε, έκθεση από κοινού με τον συνάδελφο Ανίν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του. Είναι πολύ ολοκληρωμένο το έγγραφο που αντιμετωπίζει τα βασικά προβλήματα στον τομέα των ε, βασικών μετάλλων. Βιομηχανία, βασικό μετάλλων, αλουμίνιο και χάλιβα κυρίω αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλε δυσκολίε. Είναι καιρό για αναδιάρθρωση ώστε να υπάρξει βιωσιμότητα μακροπρόθεσμα, όπως ήδη αναφέρθηκε από τον ε, συνάδελφό μου, να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο και να είμαστε κοντά στην πράσινη οικονομία. Μια από τι μεγαλύτερε προκλήσει είναι η ανάγκη να δράσουμε στον τομέα τη κλιματική αλλαγή, αλλά από την άλλη να είμαστε και οικονομικά επιτυχημένοι. Γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε οι ευρωπαϊκές πολιτικές στο κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη και καινοτομία και αλλαγή και να μην ε, περιοριστούν στην δυναμία της παραγωγής. Ένα βήμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι η μεταρρύθμιση του συστήματος ETS. Ένα άλλο θέμα που φύγει η έκθεση είναι η μείωση της ανταγωνιστικότητας ε, των βασικών μετάλλων στην Ευρώπη, στην παγκόσμια αγορά. Αυτό οφείλεται στο υψηλό κόστος της ενέργειας και στις ε, μη διοικητικές πρακτικές, εμπορικές πρακτικές, οι οποίες συμβάλλουν επίσης σε αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν σε παγκόσμιο επίπεδο να υπάρξει ισότητα, ισοτιμία όπως είπε ο κύριος Μαρτέν, παράλληλα αυτή η έκθεση αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα, πολύ ε, αποτελεσματικά, αλλά κάποια άλλα θέματα δεν θίγονται παρκώς. Θα πρέπει το ψηλό κόστος της ενέργειας να, δει στο να στο πλαίσιο της ενεργειακής έννοιας. Αυτό αποτελεί βασική προτεραιότητα των προτάσεων της Επιτροπής. Πρέπει να έχουμε μια ενιαία εσωτερική ενεργειακή αγορά που θα οδηγήσει και στην βελτίωση της κατάστασης ε, που επικρατεί στα βασικά μέταλλα, ειδικά σε σχέση με το κόστος της ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να πιέσουμε ε, να υπάρξει ένα ενεργικό κεφάλαιο ε, στο πλαίσιο του TTIP, ώστε να έχουμε Χαμηλέ τιμέ. Επίσης η ενεργειακή απόδοση πρέπει να αναφερθεί και τα προβλήματα στην ε, ζήτηση καθώ και στην επένδυση, θέματα που έχουν να κάνουν με τι δεξιότητε, την απασχόληση και η ανάπτυξη και η έρευνα. Καταλήγοντα θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό έγγραφο και ανυπομονώ να εργαστώ μαζί σα ε, σε αυτό το θέμα που αφορά τα βασικά μέταλλα της Ευρωπαϊκής Μηχανίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λόπες Βερμέχο. Καλησπέρα σας Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω τον εισηγητή εννοώ και την ομάδα του γιατί βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ θετική. Συμμεριζόμαστε ένα μεγάλο τμήμα των προτάσεων αυτών και γι' αυτό θα θέλαμε να σας συγχαρούμε. Θα ήθελα να πω επίσης ότι σημεριζόμεθα χωρίς αμφιβολία την ανάγκη που υπάρχει να συντηρήσουμε σωστά την καλλιβουργία στην Ευρώπη. Είναι στρατηγικός τομέας για την λειτουργία του βιομηχανικού τομέα και την διατήρηση ενός ευρύτατου βιομηχανικού παραγωγικού πλαισίου και η αντιστάθμιση των εισαγωγών ε, σε επίπεδο εκπομπών είναι κάτι που δημιουργεί προβλήματα στους Ευρωπαίους παραγωγούς οι οποίοι σήμερα έχουν μεγάλη υψηλή αποδοτικότητα ενεργειακή και πρέπει να διατηρήσουν τη θέση τους. Νομίζω λοιπόν ότι η δημιουργία της ισότητας είναι ο βασικός στόχος. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα θέματα τώρα στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Καταρχάς η σημασία την οποία έχει η χαλιβουργία και η βιομηχανία γενικότερα για τη συνοχή της ευρωπαϊκής οικονομίας τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται φαινόμενα μετακινήσεων των βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη για διάφορους λόγους. Γι' αυτό θα θέλαμε να υπάρξουν κάποιες προτεραιότητες όπως η αναδιατύπωση μιας πολιτικής επαϊοσύνης θα έλεγα εδώ μέσω και της χρήσης κρατικών επιδοτήσεων για να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την συνοχή των ευρωπαϊκών περιφερειών και μία επίσης συμμετοχή της Ευρώπης στην ανακαίνιση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων την επικαιροποίηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα των περιφερικών μονάδων. Το δεύτερο τμήμα αφορά την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και το κόστος της ενέργειας της ηλεκτρικής. Πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλό κόστος για το σύνολο της βιομηχανίας. Θα πρέπει να επιτροπεί στον τομέα να διαπραγματευτεί τιμολόγια ενεργειακά ε, ικανοποιητικού ε, ύψους έτσι ώστε ε, να διαφοροποιηθούμε από, τη, από τις τάσεις τις οποίες έχουμε σήμερα, ιδιαίτερα στη δική μου χώρα την Ισπανία θα πρέπει να δούμε ακριβώς ποιο είναι το μέσο κόστος της παραγωγής όπως επίσης και το λεγόμενο περιθωριακό κόστος για τα μεγαλοπόλια και τα ολιγοπόλια τα οποία κυριαρχούν. Έτσι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τους τοπικούς πόρους όπως οι ανανεώσιμες πηγές και ο άνθρακας. Νομίζω ότι αυτό ε, δεν θα πρέπει να δημιουργήσει ένα επιπλέον κόστος για τους τοπικούς τελικούς καταναλωτές. Νομίζω ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία με τον εισηγητή και θα δώσουμε την τελική μορφή στην έκθεση αυτή που είναι πολύ καλή, συμμεριζόμεστα τις θέσει της. Ευχαριστώ την κυρία Μπερνέχο. Τώρα ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο κ. Σαλίνη, αλλά συνέβη κάτι απρόβλεπτο και δεν μπορούσα να είμαι εδώ ε, για να ακούσω τον εισηγητή. Θα ήθελα σαν σκιώδης εισηγητής να κάνει κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Η πρώτη, Επαναλαμβάνω την εκτίμησή μου για τη δουλειά που έγινε μέχρι τώρα. Η δουλειά αυτή ε, έγινε και με επισκέψεις επιτόπου σε παραγωγικές περιοχές ε, του εισηγητή, κάτι το οποίο ενισχύει το περιεχόμενο της έκθεσης. Νομίζω λοιπόν ότι έχουν πλέον εντοπιστεί τα προβλήματα και οι δυσκολίες και ανοίγει η συζήτηση πάνω σε ορισμένες από τις λύσεις οι οποίες προτείνονται για να επιτευχθεί μια ρεαλιστική λύση. Ποιοι είναι οι δεσμοί αυτοί που πρέπει να ανοίξουν. Δεν θα ήθελα να μπούμε σε ε, ιδιαίτερο βάθος και λεπτομέρεια, αλλά έχουμε βασικά μια Ευρώπη η οποία είναι πολύ αποδοτική και ανταγωνιστική στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος για την επεξεργασία χάλιβα, την επεξεργασία αλουμινίου, την επεξεργασία δευτερευόντων μετάλλων. Είμαστε λοιπόν στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος σωστοί, αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε αυτά τα στοιχεία να μας οδηγήσουν σε μια διαφορετική κατάσταση, σε μια τρίτη θέση. Όταν η βιομηχανία δεσμευόμενη στον τομέα τον περιβαλλοντικό καταλήγει με ενεργειακά κόστη διόλου ανταγωνιστικά, δεν έχει λύσεις και θα πρέπει να παρέμβει στο κόστος ε, το μισθολογικό, στο κόστος του προσωπικού. Δεν είναι σωστό λοιπόν να κάνει βήματα προς τα πίσω η χαλιβουργία σε σχέση με τις κοινωνικές κατακτήσεις που δείχνουν ότι πάντα σέβεται ε, την εργασία και την έννοια της εργασίας, την ιδέα της εργασίας, θα πρέπει να μειώσουμε το κόστος της ενέργειας. Δεν πιστεύω ότι το θέμα της ρύθμισης του τιμήματος στα σύνορα είναι κάτι το οποίο είναι η μοναδική λύση για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου υπάρχει το πρόβλημα της εναρμόνισης των αντισταθμισμάτων των άμεσων μορφών κόστους. Και εγώ είμαι ανάμεσα σε αυτούς και το έχω πει επανειλημμένα που δέχομαι να υπάρξει ουσιαστική κριτική στο σύστημα του ATS το οποίο έχει πολλά στοιχεία αδυναμίας. Αλλά δεν μπορούμε να φανούμε τόσο ριζοσπάστες αγνοώντας όλα τα προβλήματα και τις σκιές οι οποίες υπάρχουν σε σχέση με την προσαρμογή των, των, του υπολογισμού των ποσοτήτων διοξίδιου του άνθρακα. Εμείς έχουμε στη χώρα μου, επειδή έχουμε μεγαλύτερες εισαγωγές από ό,τι εξαγωγές στον τομέα του διοξιδίου, κίνδυνο να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που θα κατεβάσουν το επίπεδο ανταγωνιστικότητας και ποια είναι τα benchmark αναφοράς τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να ορίσουμε τους νέους δείκτες. Ο κύριος Ταμπουράνο. Μας ικανοποιεί το ότι ακριβώς η έκθεση του Μαρτά πηγαίνει στην σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι βέβαια να δει κανεί το θέμα. Το πρώτο αφορά την εσωτερική αγορά. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις ανισότητες που δημιουργούνται στα κράτη-μέλη μέσω διαφορετικών φορολογικών πολιτικών και διαφορετικού ενεργειακού κόστους. Έτσι οι χώρες οι οποίες υφίστανται τα προβλήματα της κρίσης έχουν μεγαλύτερο δρόμο να διανύσουν. Η ρύθμιση ε, στα σύνορα όπως λέμε ε, των ποσοτήτων διοξιδίου του άνθρακα είναι κάτι το οποίο δεν οδηγεί στην ισότιμη μεταχείριση όλων των παραγωγών στην Ευρώπη. Θα πρέπει να υπάρξει ένα πρώτο βήμα λοιπόν για μια σωστή κατανομή του κόστους ανάμεσα στους Ευρωπαίους παραγωγούς και τους ε, παραγωγούς εκτός Ευρώπης. Οι ποσοστώσεις εκπομπών δεν κοστίζουν τίποτα έχει δημιουργηθεί μια, ένα απόθεμα σταθερότητας για το ATS. Η ρύθμιση λοιπόν στη, στα σύνορα ακριβώς του προβλήματος των εκπομπών δεν έχει σαν βασικό στόχο την ισότητα και την δικαιοσύνη. Θα πρέπει να δούμε ότι σαν ευρωπαϊκή βιομηχανία έχουμε υψηλά κόστη για την προστασία των εργαζομένων, το κράτος κοινωνικής προστασίας και τα λοιπά, οι οποίες είναι ε, τεκμηριωμένες βέβαια, δικαιολογημένες και από τις διεθνείς ε, οργανώσεις, τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες και τα λοιπά. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε την επερχόμενη απειλή, το TTIP, ε, να δούμε αν οι κανόνες οι οποίοι διέπουν σε κοινωνικό και παραγωγικό επίπεδο τη χαλιβουργία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αντίστοιχοι με τους δικούς μας. Θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι αλλαγές μπορούμε να κάνουμε στην, για την συμφωνία αυτή γιατί τότε θα έλεγε κανείς ότι δουλεύουμε εις είναι βασικά τα μέταλλα τα βασικά, είναι βασικά επίσης και ε, τα μέσα για τις ανανεώσιμες πηγές και θα πρέπει να εντάξουμε στον κατάλογο και τα σπάνια μέταλλα και τις σπάνιες γέες που είναι μεν σε ε, μικρό επίπεδο και σε μικρή ποσότητα αλλά παίζουν μεγάλη σημασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ε, σπάνια γέα εν πάση περιπτώσει και γι' αυτό ακριβώς ε, δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ε, παρά μόνο με τις ποσότητες των υλικών τα οποία εισάγει για να καλύψει τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές της ανάγκες. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να καλύψουμε και το θέμα της περιβαλλοντικής μόλυνσης και να προσπαθήσουμε ακόμα και μέσω της ανακύκλωσης ε, να δούμε τι θα γίνει με την εξάρτηση από τις εναλλακτικές πηγές ε, ενέργειας, μακροπρόθεσμα βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκ μέρους της EFDD ήταν ο κύριος Ταμπουράνο. Να περάσουμε τώρα στους υπόλοιπους ε, συναδέλφους ευρωβουλευτές. Ο κύριος Γκέρεκ, σας δίνω το λόγο παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα καταρχάς... Ε, ο όρος κοινά μέταλλα δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Ας πούμε ο χαλκός είναι κοινό μέταλλο, ρωτάω εγώ. Είναι ένα ημιπολίτημο μέταλλο και νομίζω ότι αυτή η υπεραπλούστευση δεν είναι πάρα Δεν μας διευκολύνει πάρα πολύ. Μιλάμε για μέταλλα τα οποία χρησιμοποιούνται ε, ως ε, μέταλλα στις κατασκευές ε, και δεν μιλάμε για μέταλλα που χρησιμοποιούνται, για λίθους ημιπολίτημους που χρησιμοποιούνται για παράδειγμα στα κοσμήματα. Τώρα είτε μιλάμε για το χάλιβα είτε για οτιδήποτε άλλο, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα μέταλλα και για την αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και για άλλες βιομηχανίες. Αν γίνει εξωτερική ανάθεση αυτό τη ε, βιομηχανία σε άλλε χώρε, ε, προφανώ αυτό δεν θα είναι επικερδέ για κανέναν τομέα τη βιομηχανία, οι, ε, οι οποίοι άλλοι τομεί μπορεί και αυτοί να φύγουν εκτό ε, Ευρώπη. Υπάρχουν ας πούμε πολύ ενεργοβόροι τομείς όπως είναι η μεταλλουργία, ε, η εξόριξη. Υπάρχουν άλλοι ε, βιομηχανικοί τομείς που είναι επίσης πολύ ενεργοβόροι. Για παράδειγμα, τσιμεντοβιομηχανία. Και ε, αυτή βρίσκεται σε μειονεκτική κατάσταση στην Ευρώπη γιατί ακριβώς απαιτεί χρήση, πολύ, μεγάλη, πολύ μεγάλη χρήση ενέργειας. αν θέλουμε να υπάρξει μια νέα εκβιομηχάνηση της Ευρώπης, για να το πω έτσι, ε, δεν είναι δυνατόν να μην είμαστε αυτόνομοι. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε στην Τουρκία, στη Μέση Ανατολή ή στην Κίνα για να αγοράζουμε ε, τα, τις πρώτες ύλες μας εκεί πέρα. γιατί στο, σε, τελική ανάλυση αυτό δημιουργεί μια εξάρτηση και αν στις πρώτες ύλες, στις στρατηγικές πρώτες ύλες έχουμε εξάρτηση από πολιτικής απόψεως είμαστε πάλι εξαρτώμενοι από άλλους ανθρώπους ανεξαρτήτως από το από ποιους το αγοράζουμε, τα αγοράζουμε. Συμφωνώ με τον εισηγητή μας ότι μία απότομη αύξηση ε, στις άδειες εκπομπών θα είναι ε, θα δημιουργήσει πρόβλημα στον ανταγωνισμό. Ναι, σε αυτό συμφωνώ. Όπως επίσης και η μετατόπιση, η μετεγκατάσταση της παραγωγής εκτός Ευρώπης θα είναι προβληματική όσον αφορά την, ε, ε τον έλεγχο, ε, στα, τον, την προσαρμογή στα σύνορα ώστε να συμπεριλαμβάνονται, ε, ώστε, ώστε στις τιμές, στον υπολογισμό των τιμών να συμπεριλαμβάνεται η πτυχή ε, της μείωσης του διοξιδίου του άνθρακα. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο το συζητήσουμε στην ε, ε, ε, κλιματική διάσκεψη που θα λάβει η χώρα στο Παρίσι σύντομα. Επίσης, πραγματικά, κυρία Μαρτέ, εγώ θαυμάζω το, το, το κουράγιο σας όταν λέτε ότι κάποια κράτη-μέλη δημιουργούν στρέβλωση ανταγωνισμού αγοράζοντας ε, ε, ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχαρητήρια που είχατε αυτό το σθένος κύριε Μαρτέ αλλά δεν υπάρχει λόγος να, το, να το θεσμοθετήσουμε και νομοθετικά αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Νίκα. Για μένα αυτή η του κύριου Μαρτέν αν θα μπορούσα να κάνω μία σύγκριση, είναι σαν τη διάγνωση ενός γιατρού που πρέπει να αποφασίσει ποια μέθοδος θεραπείας θα ακολουθηθεί και ποια όχι. Αυτή η έκθεση και πρέπει να πω ότι εργάστηκε εξαιρετικά ο κύριος Μαρτέν. Βρίσκει κανείς αυτά τα στοιχεία. Είμαστε θύματα αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Αφενός είναι πολύ σημαντικό οι εκτιμήσεις αντικτύπου να μην ε, εκτελούνται τόσο σχολαστικά. Πρέπει να δούμε ποιες ε, θα είναι οι τιμές στην ενέργεια από το περιορισμό των εκπομπών του διοξείου του άνθρακα. Αν, παραδείγματο χάρη, θα είναι πολύ ψηλέ οι τιμές σε έτοιμα προϊόντα από ε, την χαλιβουργία και από την βιομηχανία του αλουμινίου. Αν ανεβούν οι τιμές, τότε αυτό θα οδηγήσει στην ε, μείωση της ανταγωνιστικότητας αυτών των βιομηχανιών. Κάτι που πρέπει επίσης να το αποκλείσουμε. Κάποιοι ίσως να χαίρονται ε, με μέτρα που θα οδηγήσουν σε ένα πιο καθαρό αέρα, σε καθαρή ατμόσφαιρα, αλλά κάποιος πρέπει παρόλα αυτά να παράγει αλουμίνιο και χάλιβα στην Ευρώπη. Ειδικά όταν κάποιες χώρες ε, εκτός Ευρώπης είναι υπεύθυνες για πάνω από 5% των εκπομπών άνθρακα. Η πολιτική αυτή λοιπόν είναι κάπως ασυνεπής, δεν έχει συνέχεια και πολύ σπάνια βλέπουμε να υπάρχει ξεκάθαρη τοποθέτηση και από την πλευρά της Επιτροπής. Ε, το αφήνουμε στη θέληση του Θεού. Αν έχουμε τύχη μπορεί να, να το πετύχουμε, ίσως και όχι. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε και να, να κατανοήσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό κλάδο η χαλιβουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν στρατηγική σημασία αυτά τα υλικά και θα είναι πάντα απαραίτητα. Δεν μπορούμε να τα εισάγουμε επαόριστο. Και αν δεν είμαστε πλέον ανταγωνιστικοί και πρέπει να εισάγουμε αυτά τα υλικά, ίσως θα πρέπει να αποφασίσουμε να σταματήσουμε να παράγουμε, όμως αυτό θα έχει πολύ ψηλό κόστος. Αν θέλουμε μια ανταγωνιστική βιομηχανία, θα πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρχουν ε, όλες τις περισσότερες αυξήσεις στην εφορολόγηση Ε, υπό το φως και το, το πνεύμα των ε, περιβαλλοντικών στόχων. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι δικό μας έργο στην Επιτροπή Ήτρε να αναλάβουμε δράση όταν επεξεργαζόμαστε αυτά τα θέματα στους φαγγέλους πρέπει να προσέχουμε ότι τα θέματα αυτά έρχονται και σε εμάς και δεν τα ε, ε, διαχειρίζεται μονάχα η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι και για την βιομηχανία και για ό,τι έχει να κάνει με την βιομηχανία. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα. Μέθοδοι. Ε, ναι, θα σας παρακαλέσω να, είστε, να κρατάτε το χρονικό όριο. Όλοι μιλάνε για 20 το παραπάνω. Κυρία Ρόζα Νταμάτο, τρία λεπτά σας παρακαλώ. Και συγγνώμη που ξεκινάω από εσάς που είστε μια κυρία. Θα ήθελα δύο σημεία να θέσω. Να υπογραμμίσω καταρχάς ότι τίθεται το θέμα του σεβασμού του περιβάλλοντος και των ουσιών που μολύνουν το περιβάλλον και δεν αναφέρουμε μόνο στο διοξίδιο του άνθρακα. όλες οι υπάρχουσες χαλιβοργίες θα πρέπει να σέβονται συγκεκριμένους κανόνες και οι ευρωπαϊκές. Οι εγκαταστάσεις αυτές επηρεάζουν ιδιαιτέρως την υγεία των εργαζομένων αλλά και γενικότερα των πολιτών που ζουν σε γειτονικέ περιοχές. Και είναι σημαντικές οι μονάδες αυτές και για άλλες βιομηχανίες όπως ο τουρισμός, η γεωργία, η κτηνοτροφία κτλ θα πρέπει να καταλήξουν σε μία λύση θα έλεγα δραστική αν οι εγκαταστάσεις είναι αντιοικονομικές και ξεπερασμένες και παραμένει σε λειτουργία η μονάδα μόνο ε, χάρη στις κρατικές επιδοτήσεις. Θα ήθελα να μάθω αν αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να αλλάξει το πρότυπο ανάπτυξης, να δείξει θάρρος και να μην έχει στόχο μόνο σε μια απλή αύξηση της κατανάλωσης, μια αύξηση του κύκλου εργασιών του εμπορίου, της παραγωγής και κατανάλωση κατανάλωσης αναπόφευκτης των φυσικών πόρων. Θα πρέπει να επανέλθουμε όπως λέει ο εισηγητής και στα θέματα των ε, εναλλακτικών πηγών αλλά με διαφορετική η αντίληψη, όχι με συγκεντρωτικές αντιλήψεις, με τεράστιες εγκαταστάσεις, α, με ολική ή ελιακή ενέργεια. Και υπάρχει φυσικά και το θέμα της αποδοτικότητας, της ενεργειακής. Θα πρέπει να υπάρξει μια νέα οικονομία, μια οικονομία η οποία να είναι κοντά σε αυτήν την ευλογημένη θα έλεγα κυκλική οικονομία να παράγουμε λιγότερο και να προχωρήσουμε σε μια οικονομία ανακατανομής βγαίνοντας επιτέλους από τη δεύτερη βιομηχανική επανάσταση και αγκαλιάζοντας την τρίτη βιομηχανική πλέον επανάσταση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά και το περιεχόμενο όσων είπατε, αλλά ήσασταν και πάρα πολύ σύντομοι. Η κυρία Δελκαστίο. Uh, λοιπόν, να τα πω στα ισπανικά. Θέλω να ευχαριστήσω τον Εντουάρδο Μαρτίν για την πρότασή του. Είχαμε την δυνατότητα να τα συζητήσουμε αυτά είναι σαφής η πρότασή σου, είναι συγκεκριμένη και συνοπτική. Αυτό το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα επί της ουσίας. Έχω δύο ερωτήσεις μόνο να θέσω. Η μία αφορά το θέμα της ρύθμισης στα σύνορα. Των ρυθμίσεων λοιπόν στα σύνορα για το διοξίδιο του άνθρακα Υπάρχουν εδώ δύο διαφορετικά προβλήματα, τουλάχιστον έτσι το βλέπουν οι επιστήμονες. Ε, είναι το θέμα των έμεσων εκπομπών και εκεί υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί γιατί είναι δύσκολο σε επίπεδο ε, διοικητικό αν θέλετε, διαχειριστικό να υπολογίσει κανείς το ενεργειακό κόστος και τίμημα στις εισαγωγές. Ε, θα χρησιμοποιεί γι' αυτό τον μηχανισμό της χώρας παραγωγής ή κάποιον άλλο μηχανισμό καθορισμού της τιμής. Ενώ για τις άμεσες εκπομπές τα πράγματα είναι πιο εύκολα, είναι πιο ε, απλά. Θα μπορούσε λοιπόν να υπάρξει μια τέτοια λειτουργία σε επίπεδο εναρμονισμού του κόστους. Ε, πάνω σε όλα αυτά ισχύει και η ανάγκη που υπάρχει ε, με συμβάσεις ε, μικρής διάρκειας. Νομίζω ότι οι μακροπρόθεμες συμβάσεις με εναρμονισμένα κριτήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα κρίσιμο σημείο για την βιομηχανία και του αλουμινίου και του χάλιβα. Σας τα θέτω λοιπόν και περιμένω τις απόψεις διαφορά δηλαδή που υπάρχει ανάμεσα στις άμεσες και έμεσες εκπομπές και τη ρύθμιση στα σύνορα και πώς η μία λειτουργεί εις βάρος ή υπέρ της άλλης. Um, Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφε Ντελεκαστήγιο. Να ζητήσουμε κάποια σχόλια τώρα από την κυρία Μάτια Πελεγκρίνη. Πάνω στο ίδιο θέμα, παρακαλώ. Δεν είμαι κύριο, κυρία, με συγχωρείτε, είμαι κύριος. Δεν ήταν επακριβής η ενημέρωσή μου, είναι ο κύριος της Επιτροπής και όχι η κυρία της Επιτροπής. Θα είμαι σύντομος. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ενδιάμεση έκθεσή του. Ήδη είχαμε την δυνατότητα να συζητήσουμε την πρώτη πρόταση σε άλλη ημερομηνία. Νομίζω ότι η πρόκληση η οποία έχει εντοπιστεί από διάφορες κοινοβουλευτικές τροπολογίες είναι γνωστές οι τροπολογίες αυτές. Εμείς έχουμε μια μεγάλη εξάρτηση για τη βιομηχανία σαν παράδειγμα των, uh, των βηματοδοτών. Ε, έχουμε επίσης και στα βασικά μέταλλα και στις σπάνιες και στα σπάνια μέταλλα έχουμε μείνει πίσω γενικά. Αυτός είναι και ο λόγος λοιπόν για τον οποίο πολλοί από σας είπατε ότι απαιτείται μια πολιτικής συνοχής. Απαιτείται να συνδυάσουμε από τη μία τον αγώνα κατά της, ε, των κλιματολογικών συνεπειών και από την άλλη να διατηρήσουμε το επίπεδο της βιομηχανίας ιδιαίτερως ανταγωνιστικό. Έχουμε ανάγκη και από την παραγωγή πρωτογενών ε, πρωτονυλών μάλλον και άκουσα αυτά που είπατε για την κυκλική οικονομία. Ξέρετε ότι εμείς θα προτείνουμε ένα νέο πακέτο κυκλικής οικονομίας μέχρι το τέλος του χρόνου. Αλλά αυτή από μόνη δεν μπορεί να βοηθήσει. Αν δείτε σαν παράδειγμα την ανακύκλωση ε, χαλκού στην Ευρώπη δεν ικανοποιεί ούτε το 30% της ζήτησης και ακόμα και αν αυξηθεί η δυνατότητα αυτή πάλι δεν θα καλύψουμε τις ανάγκες. Απαιτείται λοιπόν να προχωρήσουμε και σε σχέση με την ανακύκλωση και σε σχέση με την πρωτογονή παραγωγή. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίσει η βιομηχανία αυτή, ιδιαίτερα σε σχέση με τον προϋπολογισμό για την ενέργεια. Εμείς στην Ευρώπη έχουμε μια κατάσταση ε, η οποία δεν αφήνει να προχωρούμε σε μακροπρόθεσμες συμβάσεις και γι' αυτό θα πρέπει μέσω της Ένωσης για την Ενέργεια, της Ενεργειακής Ένωσης να αναζητήσουμε νέες λύσεις. Να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά εσάς και τον εισηγητή ε, να πω ότι αυτά τα οποία είπατε για τη μεταρρύθμιση των ATS θα ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παλεγκρίνη. Τμήματάρχης της, ε, για στη Γενική Διεύθυνση ε, Ανάπτυξης που μόλις δημιουργήθηκε. Κύριε Σιγητά, ακούσατε πολλά θετικά σχόλια. Ποια είναι η άποψή σας. Πράγματι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους ε, που έλαβαν το λόγο. Δεν θα μπορέσω να απαντήσω στο σύνολο των ερωτήσεων. Ε, ε, μόλις άρχισε η εργασία μας, θα υπάρξουν συναντήσεις με τους κοιόδης εισηγητές, θα υπάρξουν τροπολογίες, θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το κείμενο και να λάβουμε υπόψη ως το δυνατόν περισσότερες παρατηρήσεις. Τώρα, περί τίνος πρόκειται. Παρά ε, τις ε, ε, ιδέες που μπορούμε να έχουμε στο μυαλό μας ε, υπάρχει σε γενικές γραμμές σε παγκόσμιο επίπεδο αύξουσα παραγωγή ενώ είναι ευθύνουσα στην Ευρώπη δεν λέμε ότι ξαφνικά ε, θα πάμε ε, στους 250-300 εκατομμύρια τόνους ατσάλι το χρόνο αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε να κάνουμε αυτή την επιλογή ή θα πάμε σε μια θα, θα μεταφέρουμε την παραγωγή μας σε άλλες υπήρους που δεν σέβονται ε, τα πρότυπά μας ε, τα πρότυπά μας τα περιβαλλοντικά ούτε δημόσια υγεία ή θα παραμείνει η παραγωγή στην Ευρώπη αλλά ε, ε, τουλάχιστον εδώ έχουμε, είμαστε υποδειγματικοί ως προς τις προδιαγραφές που θέτουμε για, τις, για, για, τον σεβασμό του περιβάλλοντος. εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να διαλέξουμε μεταξύ της υγείας και της παραγωγής στη συγκεκριμένη έκθεση. Μπορούμε να έχουμε μια καθαρή παραγωγή σεβόμενη το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Και όταν μια επιχείρηση δεν το κάνει αυτό, πρέπει να υφίσταται όσοι, γιατί η νομοθεσία το επιτρέπει αυτό. Τώρα, για όλα τα υπόλοιπα, για την προσαρμογή στα σύνορα. Αυτό μας το είπαν οι τοπικοί παράγοντες επιχειρηματίες. Αυτό που τους, ε, ε, τους τρομάζει πάρα πολύ είναι αυτή η πολιτική ε, ETS και σας το λέω αυτό για να σας εξηγήσω ότι όταν πήγαμε στον Ντίσελντορφ στην Γερμανία, επειδή μιλάμε ε, με τον... Ε, με, με, και μιλούσαμε με τους, επιχειρηματο με τους επιχειρηματίες εκεί, ε, μας είπε ε, μας είπαν ότι αυτά τα 150 εκατομμύρια θα τα επενδύσω εκτός Ευρώπης γιατί εκεί δεν θα μου δημιουργήσουν επιπλέον προβλήματα και δεν θα μου θέσουν επιπλέον περιορισμούς. Αυτό λοιπόν το ε, επιπλέον κόστος του διοξιδίου του άνθρακα πώς θα το αντιμετωπίσουμε και το γεγονός ότι μετακυλίεται στον ε, πελάτη. Πρέπει να υπάρχει μια ισότιμη μεταχείριση στην προκειμένη περίπτωση με, το, με την Κίνα. Αν μπορέσετε να το κάνετε αυτό, εγώ αυτά τα 150 εκατομμύρια θα επενδύσω στην Κίνα, αλλά στην Ευρώπη. Αυτή τη δυσκολία έχουμε σήμερα. Γιατί α δούμε τα, νούμερα. Ακόμη κι αν είμαστε οι καλύτεροι, η Ευρώπη, η σιδηρουργία για παράδειγμα, ρηπαίνει σήμερα περισσότερο από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Γιατί δεν υπάρχουν επενδύσει. Οι επενδύσει είναι αυτέ που μα λείπουν. Η έλλειψη ανταγωνιστικότητας, η έλλειψη σεβασμού περιβάλλοντος ε, υπάρχουν επειδή υπάρχει αβεβαιότητα της πολιτικής ETS ε, ε, και δεν υπάρχουν επενδύσεις. Λοιπόν, ε, το, το επιπλέον ε, που θέλουμε να ε, επενδύσουμε πρέπει να πάει στις τσέπες των δικών μας των επιχειρηματιών και των βιομηχάνων και, παράλληλα να συνεχίσουμε να σεβόμαστε την, το, το περιβάλλον με λιγότερη ατμοσφαιρική μόλυνση και την επίτευξη όλων των υπολείπων στόχων μας έχουμε να περάσουμε, θέλουμε να περάσουμε σε έναν ενάρετο ε, κύκλο, θέλουμε να τους πούμε ε, στους βιομηχάνους μας ότι θα τους βρούμε έναν τρόπο χρηματοδότησης και να πούμε, να δώσουμε ένα, ένα μήνυμα στους εκτός Ευρώπης ότι αν θέλετε να επενδύσετε στη δική μας την Ήπειρο θα πρέπει να σέβεστε τις προδιαγραφές μας. Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι απλώς ο μεγάλος αφελής ε, της υπόθεσης. Η είναι παγκόσμιος ο ανταγωνισμός και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό. Όσον αφορά τη δυσκολία των μακροπρόθεσμων ε, ε, συμβάσεων, ναι, υπάρχουν και σε άλλε χώρε. Μα το λένε αυτό παρά το γεγονό ότι το κόστο ε, των επενδύσεων είναι μεγάλο. Αυτό που του επασχολεί είναι το η έλλειψη της ορατότητας. Δεν μπορούμε σήμερα να, δεν μπορεί να, σήμερα να ε, πληρώσει, να, να δώσει ένα χι ποσό για μια συγκεκριμένη σύμφω, ε, ε, σύμβαση ηλεκτρισμού για παράδειγμα και να το αντικαταστήσει αυτό με ένα συμβόλαιο 10-15 ετών χωρίς τις απαραίτητες επενδύσεις. Και υπάρχουν και άλλα, υπήρξαν πολλά άλλα ερωτήματα σχετικά με το θέμα αυτό και τι θέλω να πω ότι η δική μας διάγνωση βρίσκει τους πάντες σύμφωνους. Αυτούς τους τέσσερις πυλώνες που ε, θεωρούμε ε, ότι υπάρχουν είναι οι τοπικοί, τοπικός, ε, οι τοπικοί παράγοντες, είναι οι επιχειρήσεις, είναι οι βιομήχανοι και είναι και οι ε, τοπικοί εκπρόσωποι. Αυτό θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης με σεβασμό του περιβάλλοντος, με σεβασμό της δημόσιας υγείας και παράλληλα να στείλουμε και ένα ισχυρό μήνυμα προς τα έξω. Και νομίζω ότι αυτή η έκθεση με όλα αυτά που υπόθηκαν δεν θα μπορεί παρά να είναι ένα πολύ καλό σημείο αφετηρίας. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ. ευχαριστώ για τις απαντήσεις, για τις παρατηρήσεις. Και τώρα και στην εισαγωγική ομιλία και τώρα να πω ότι προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών είναι η 3η Ιουλίου του 2015, 12 η ώρα το μεσημέρι. 3 Ιουλίου. και θα εκταστούν οι τροπολογίες την 3η Σεπτεμβρίου, δύο μήνες δηλαδή, από τις διακοπές. Σας ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή, όλους τους συναδέλφους για τη συζήτηση και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα περάσουμε στο σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης. Οργανισμός Εργασίας Εθνιστικών Ορχών Ενέργειας, ACER, το Συμβούλιο των Ρυθμιστών και η ACER εκπροσωπούνται εδώ. Είναι εδώ μαζί μας. John. John okay. Okay. There's no, no visible sign that you are together with us. They're coming. Coming. Coming. Immediately. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ σημαντικό σημείο. Ανταλλαγή απόψεων. Στον Αλβέρντο Ποτότσνικ, διευθυντή του ΆΣΕΡ, του Οργανισμού Συνεργασίας Ερθμιστικών Αρχών Ενέργειας, Ιταλός. Κύριος Ποτότσνικ, η Σλοβενία και τα είναι πολύ κοντά η μία στην άλλη. Λοιπόν, ευχαριστώ. Και ο κύριος Λότμοργ, πρόεδρος του Συμβουλίου της Άσερ των Ρυθμιστικών Αρχών. Η συζήτηση αφορά ένα πολύ σημαντικό θέμα, το σχέδιο προγράμματος εργασίας του Άσερ το 2016. Θα συζητήσουμε το θέμα αυτό και έχουμε ανώτατους προσκεκλημένους εδώ μαζί μας και αυτό το σχέδιο εργασιών θα πρέπει να υποβληθεί στο Συμβούλιο των Ρυθμιστικών Αρχών όπως προτείνεται από τον οργανισμό, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μέχρι τις 30 Ιουνίου, δηλαδή σε δύο εβδομάδες. Επομένως δεν έχουμε πολύ χρόνο. Γι' αυτό είναι και πολύ κρίσιμη η συζήτηση που θα κάνουμε εδώ. Να σας υπενθυμίσω στον σε κάθε επιτροπή και δύο προσκεκλημένοι είναι ευπρόσδεκτοι να επαναλάβω και όπως είναι προφανές οι τελευταίες συζητήσεις ως, ως προς την έλλειψη ανθρώπινων πόρων του ΆΣΕΡ είναι κάτι πολύ σημαντικό και αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης τον Μάια στην Ολομέλεια. Ως πρόεδρος της ΙΤΕΡ έστειλα μια επιστολή στον Άρια Σκανιέτε και στον Σεφτσοβιτς για την έλλειψη πόρων και ανθρωπίνου δυναμικού που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του οργανισμού του Άσερ. Τελευταία δήλωση της Επιτροπής για τον προπολογισμό του 2016 δημοσιεύτηκε τέλη Μαΐου και υπάρχει μια ελάχιστη αύξηση στον προπολογισμό του ΆΣΕΡ. Είναι ίσως για να εκπληρώσετε την τη θητεία σας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Διευθυντά, δεν θεωρώ ότι είναι επαρκής για να παρακολουθήσουμε παρκώς την αγορά ε, ενέργειας. Είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά σας για την εσωτερική ενεργειακή ένωση και στο αέριο και στον ηλεκτρισμό. Ασχολήθηκε με τα δύο, κάτι που δεν είναι εύκολο. Φυσικά τα διχωρίσουμε στο διάλογό μας, αλλά όλα τα προβλήματα και στους δύο τομείς είναι παρόμοιοι και αν δεν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την εσωτερική ενεργειακή αγορά, δεν θα μπορέσουμε να ε, είμαστε ασφαλείς ως προς την ενεργειακή επάρκεια. Να μειώσουμε το κόστος της ενέργειας, γιατί αυτό είναι ο στόχος μας. Και πρέπει να προηγηθεί τη θέση σε ισχύ του TTIP. Μια παρουσίαση στην αρχή, κύριε Διευθυντά, γιατί προτείνετε εσείς αυτό το πρόγραμμα εργασιών και το παρουσιάσετε και στο ε, Συμβούλιο των Διευθυντών. Να θέξετε λοιπόν τα πιο σημαντικά στοιχεία. Ο λόγος εσάς παρακαλώ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να είμαι μαζί σας σήμερα. Σας ευχαριστώ και για την υποστήριξη που το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σας έχει προσφέρει στην υπηρεσία από τότε που δημιουργήθηκε. Την πρώτη φορά που ήρθα εδώ ήταν το 2010. Ο Λόντ Μόρ και εγώ εκτιμούμε το πλαίσιο του προγράμματος το οποίο σας υποβάλαμε ή μάλλον θα υποβάλουμε στο τέλος του μήνα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Κοινοβούλιο και στην Διευθυντική Επιτροπή. Στο τέλος του χρόνου θα εγκριθεί από την Διευθυντική Επιτροπή και θα ακολουθήσει η έγκριση της Διοικητικής Επιτροπής. Εκτιμούμε την δυνατότητα που έχουμε να συλλέξουμε τις αντιδράσεις και τις ιδέες σας έτσι ώστε να αντιλάβουμε υπόψη μας για την τελική μορφή του κειμένου μας. Πριν εγκριθεί από τις δύο επόμενες επιτροπές και πριν υπάρξει και η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμα εργασίας συνεχίζεται για φέτος περιλαμβάνοντας ε, μια πολυετή έποψη γενικά των εργασιών μας, δίνει μια μακροπρόθεσμη αντίληψη για το τι κάνει η Επιτροπή. Το πρόγραμμα αυτό θα σας το στείλουμε σε λίγες μέρες στο Κοινοβούλιο. Θα έχετε λοιπόν μια τέτοια πολυετή πρόβλεψη ε, για το μέλλον όπως το κάναμε και πέρυσι γιατί συνεχίζουμε ακριβώς την προσπάθεια να πετύχουμε τους ίδιους στόχους η πρόκληση αυτή τη στιγμή είναι να τηρήσουμε την εντολή μας με, τις λίγες, με τους λίγους πόρους που έχουμε πλέον στην διάθεσή μας. Και το πρόγραμμα το οποίο θα σας παρουσιάσουμε στο τέλος του μήνα βασίζεται στην πρόβλεψη κόστους η οποία συμφωνήθηκε το Μάρτιο με τη Διευθυντική και τη Διοικητική Επιτροπή επί τη βάση των πιστώσεων που είναι διαθέσιμες για την υπηρεσία. Δηλαδή και σε σχέση με τη διαφάνεια της αγοράς ενέργειας είναι ένα και το πακέτο υποδομών. Η προσπάθειά μας εντάσσεται ακριβώς στα πλαίσια της ενεργειακής στρατηγικής της ε, Ένωσης για την Ενέργεια νομίζω ότι επηρεάζουμε ε, με την εργασία μας τα θέματα αυτά. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στα θέματα της ολοκλήρωσης της ε, αγοράς ενέργειας και δεύτερον στο θέμα της διασφάλισης της ε, προμήθειας μετά από τα stress test τα οποία έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα στον τομέα της ασφάλειας των προμηθειών μας μέσω στενότερης συνεργασίας. Το πρόγραμμα εργασίας μας βασίζεται σε τέσσερα θεματικούς άξονες. Αυτό ίσχυσε και φέτος και υπάρχει συνέχεια στην προσπάθεια την οποία κάνουμε. Το πρώτο θέμα είναι αυτό το οποίο ονομάζονται, ε, η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Αυτός ήταν στόχος για το τέλος του προηγούμενου χρόνου. Αλλά ήμασταν μόνο στην πρώτη φάση της δημιουργίας μιας τέτοιας αγοράς. Τώρα θα πρέπει να εφαρμόσουμε και να παρακολουθήσουμε σωστότερα την εφαρμογή των ρυθμίσεων. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι το τρίτο πακέτο θα μεταφερθεί πλήρως σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας και θα πρέπει επίσης να εφαρμόσουμε σωστά και τις κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες έχουν υιοθετηθεί στον τομέα του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου. Έχουμε τα θέματα του REMIT, διαφάνεια, ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στο τέλος του 11 με την υιοθέτηση και τη θέση σε ισχύ των εφαρμοστικών πράξεων στις αρχές του 2015 η ημερομηνία για το νέο πλαίσιο ελέγχου καθορίστηκε για τον Οκτώβριο του 2015. Από τον Οκτώβριο του 2015 θα ζωντανέψει το REMIT. Θα υπάρξει μια υπεχρέωση δηλαδή όλων των συμμετεχόντων στην αγορά να τροφοδοτούν την υπηρεσία και θα μπορεί ελπίζουμε η υπηρεσία να ελέγχει την ακεραιότητα των αγορών αυτών. Υπάρχουν προβλήματα και σε επίπεδο υποδομών. Εδώ εργαζόμαστε στα πλαίσια της εντολής του τρίτου πακέτου υποδομών και συνεισφέρομαι ακριβώς και στην προσπάθεια για το δεκαετές πλαίσιο, εμπλεκόμεθα όμως και στην διαδικασία για την επιλογή και την εφαρμογή του προγράμματος κοινού ενδιαφέροντος. Εμπλεκόμεθα επίσης και στα θέματα κόστους, εκεί όπου δεν υπάρχει δυνατότητα συμφωνίας ανάμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες διαφορετικών χωρών. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε επίσης και κάποιες προκλήσεις σε σχέση με την πρωτοβουλία 2020, τι προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα 10 χρόνια και τι ρυθμιστικού τύπου απαντήσεις μπορούμε να δώσουμε. Σχετικά τώρα με την διαχείριση της αγοράς για μετά το 2014, νομίζω ότι θα πρέπει απλά να προχωρήσουμε στην εφαρμογή των κανόνων τους, τις οποίους έχουμε ήδη αποφασίσει. Στον τομέα του ηλεκτρισμού υπάρχει δυνατότητα για την εναρμόνιση της μετάδοσης όπως επίσης και για τη δομή των τιμολογίων. Παραλλήλα με την εφαρμογή αυτών των ε, κανόνων και των δομών εργαζόμαστε και με την πρώτη τροπολόγηση του πρώτου δικτύου μηχανισμού ε, κατανομής στον τομέα της αυξητικής πλέον ε, η χωρητικότητας. Πέρα από τους κανόνες απαιτείται όμως πρόοδος και μπορούμε να σας δείξουμε αυτή τη διαφάνεια η οποία σας δείχνει το τι υπάρχει ακριβώς στον τομέα της αγοράς. Ήδη μέχρι τώρα ένα μεγάλο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνεται σε μια ενιαία αγορά με μία πλατφόρμα ε, και για τον καθορισμό των τιμών και για την διακίνηση από τη Βλαρτάρ μέχρι τη θάλασσα του Μπάρεντς υπάρχει μια ε, ενιαία αγορά. Υπάρχει ένα άλλο τμήμα στην Ανατολική Ευρώπη και αυτό είναι διαδικτυωμένο έχει σίζευθεί δηλαδή, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Στο φυσικό αέριο έχει υπάρξει κάποια πρόοδος εδώ για την κατανομή της χωρητικότητας. Έχουμε μεγάλα προγράμματα, ένα μεγάλο πρόγραμμα και κάποια επιμέρους. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει χωροτεκτική πρόοδος αλλά υπάρχει επίσης και υπάρχουν και άλλα βήματα τα οποία λειτουργούν θετικά για τον καταναλωτή. Για το δεύτερο θέμα, το REMIT, έχουν τέσσερις μήνες ακόμα μέχρι τη θέση σε λειτουργία στις 7 Οκτωβρίου. Από τις 7 Οκτωβρίου και μετά οι συμμετέχοντες στην αγορά που εμπορεύονται προϊόντα, τα οποία εμπορεύονται σε οργανωμένους χώρους, Ε, θα υπάρχει η καταγραφή αυτών των δραστηριοτήτων και ελπίζουμε ότι θα ε, φτάσουμε στην καταγραφή προϊόντων που θα ισοδυναμούν σε πάρα πολύ υψηλές ποσότητες. Η σημασία του REMIT δεν χρειάζεται να υπογραμμιστεί. Να σας δώσω εδώ τα τελευταία στατιστικά στοιχεία των δραστηριοτήτων μας από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ το REMIT γιατί όπως είπα θα λειτουργήσει από τον Οκτώβριο, αλλά έχουμε ήδη αρκετές τέτοιες περιπτώσεις στην υπηρεσία. 67 τέτοιες υποθέσεις έχουν διακοινωθεί, 26 έχουν κλείσει, οι 41 είναι σε εκκρεμότητα. Από αυτές που κλείσανε σε 6 περιπτώσεις υπήρξε μια παραβίαση των υποχρεώσεων στα πλαίσια του REMIT, δεν σημαίνει ότι αν ένα τμήμα της εμπορίας της ενέργειας έχει συστηματικό πρόβλημα. Αλλά αυτό δείχνει όμως ότι απαιτείται μεγαλύτερη ακεραιότητα και μεγαλύτερη διαφάνεια. Έχει γίνει πολλή δουλειά ανάμεσα στις ρυθμιστικές αρχές και την υπηρεσία έτσι ώστε το REMIT, γιατί το REMIT είναι μοιρασμένη αρμοδιότητα, Ξεκινήσαμε μια ιστο, ε, ε, ιστοθύρα, ένα πόρταλ, το Acer Remit Portal έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητες επεξεργασίας και σε επίπεδο υπηρεσίας και σε επίπεδο ε, κρατών μελών για την σωστή εκπαίδευση. Η πρόκληση στην περίπτωση αυτή όπως και σε άλλες περιπτώσεις είναι βέβαια ο προϋπολογισμός. Όπως είπα ότι το πρόγραμμα εργασίας βασίζεται στις προβλέψεις που έγιναν από την Διοικητική Επιτροπή και φτάνουν τα 20 εκατομμύρια για τον επόμενο χρόνο. Περιλαμβάνει επίσης 44 ε, υπαλλήλους και κάποια ε, ποσά για κάποια επιμέρους ε, συμβόλια, συμβάσεις μάλλον. Επί τη βάση των στοιχείων τα οποία ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγιναν προτάσεις για την ε, ε, υπηρεσία να βρεθούν άλλοι 10 υπάλληλοι με 15 επιπλέον εκατομμύρια ε, στον προϋπολογισμό. Αυτό είναι καλό. Είμαστε ευγνώμονες προς την Επιτροπή και αναγνωρίζει η Επιτροπή ότι οι πόροι τους οποίους έχει η υπηρεσία δεν είναι επαρκής για την περαιτέρω λειτουργία της αν και ακόμα και με αυτούς τους 15 είμαστε μακράν αυτού του οποίου θα επιθυμούσαμε σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού για την αναλυτική και πρακτική μας επεξεργασία προτάσεων. Θα ζητήσω τώρα, αν μου επιτρέπετε, από τον Λόρδ Μόγκ να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ευχαριστούμε κόσμο. Θα ήθελα και εγώ να ε, σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Εγώ μια διαφάνεια θα σας δείξω και θα ήθελα απλώς ε, να σας προειδοποιήσω για κάτι το οποίο μπορεί να μην δημιουργήσει δυσκολία, αλλά κατά την άποψή μας υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τη φύση του ε, Remit λόγω μιας τεχνικής ετροποποίησης, η οποία δεν έχει αυτή την πρόθεση αλλά θα έχει αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, προσπαθώ μέσω της διαφάνειας να σας το δείξω εντάχει. Δεν θα μπω σε πάρα πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά ουσιαστικά οι τρέχουσες διατάξεις ε, δίνουν στο ρέμι τη δυνατότητα χειρισμού ε, της εμπορίας της ενέργειας ε, τρία λεπτά κάθε χρόνο από ε, μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο οικονομικό πρόγραμμα και μια ολόκληρη οικονομική πολιτική δεν είναι δηλαδή ε, κάτι το οποίο δίνει τη δυνατότητα ε, στις εταιρείες να προβλέψουν το μέλλον και να κάνουν τις απαραίτητους διακανονισμούς. Αυτό λοιπόν που προτείνεται είναι μια αλλαγή. Μια αλλαγή αυτή τη στιγμή η, η επέκταση των ε, του ορισμού των οικονομικών μέσων που μπορεί να είχε ως αποτέλεσμα ε, τη μείωση των ε, ε, παρεκκλήσεων και αυτό μπορούσε να σημαίνει ότι το REMIT δεν θα αποτελεί τμήμα των επιχειρηματικών συναλλαγών των περισσότερων εταιριών γιατί ακριβώς θα γινόταν μετατόπιση πολλών διακανονισμών σε ε, ε, διμερείς ε, συμφωνίες και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εμείς είχαμε πάρα πολλές επαφές, ήρθα σε επαφή με τον Επίτροπο Χίλ και με πολλούς διευθυντές. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι θα μπορέσει ο Επίτροπος να βρει τρόπο να αποφύγει αυτές τις συνέπειες. Επειδή όμως είχαμε πάρα πολύ καλές, έχουμε πολύ καλές ε, ε, ε, σχέσεις με το Κοινοβούλιο, πιστεύω ότι πρέπει να σας προειδοποιήσω για τη ζημιά που θα μπορούσε να γίνει στις προτάσεις για το Ρέμιτα αν όντως περάσουν όλες αυτές οι προτάσεις. Αυτό βέβαια δεν θα αρχίσει πριν από το 2017 και δυστυχώς αυτή τη στιγμή λαμβάνονται οι αποφάσεις τώρα κατά τους ερχόμενους μήνες. Οπότε Μπορεί να χρειαστεί να ξαναέρθουμε να ζητήσουμε τη βοήθειά σας. Για την ώρα πάντως αυτά έχω να πω. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Ε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους ε, συναδέλφους ευρωβουλευτές. Υπάρχει μια ομάδα επαφών ε, με την ε, Acer, η κυρία Βέρνε, ο κύριος Σιλικιώτης ε, συμμετέχουν. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι. μπορείτε να λάβετε το λόγο αν θέλετε. Τι λέτε. Η κυρία Κάλλας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις έχω. Είπατε πολλές φορές ότι ο προϋπολογισμός σας δεν επαρκεί. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι για άλλα εργαλεία ή άλλες αρμοδιότητες που θα θέλατε να έχετε στη διάθεσή σας ε, για να ανοίξετε την ενεργειακή αγορά και επίσης ποια είναι η συμμετοχή του Acer ε, στον ε, σχεδιασμό, της, στον προγραμματισμό της αγοράς ηλεκτρισμού. Η κυρία Ντυρκούνεν. Ευχαριστώ πολύ παρόμοια είναι και η δική μου ερώτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν θέλουμε να έχουμε μη, έναν ε, ισχυρότερο ε, ρυθμιστή στην Ευρώπη αντί για 28 διαφορετικές ρυθμιστικές αρχές, είναι θέμα χρημάτων ή είναι θέμα νομοθεσίας. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να σας βοηθήσουμε ώστε να υπάρχει καλύτερη ρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι ισχυρότερη αυτή η μία ρυθμιστική ε, αρχή ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, εμένα ε, η ερώτηση μου και μάλλον την τοποθέτησή μου κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από τη της προηγούμενου συναδερφού, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη ότι γίνεται μια προσπάθεια να ενισχυθούν οι διασυνδέσεις, η διαφοροποίηση των πηγών και των οδών προμήθειας της ενέργειας, να δημιουργηθεί ενιαία ενεργειακή αγορά. Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς μπορεί να συμβάλλει ε, και ο Acer ώστε να τερματιστεί ή να αρθεί η απομόνωση κρατών μελών και περιοχών από τα μεγάλα ε, ηλεκτρικά και ενεργειακά δίκτυα. Δηλαδή προσπαθούμε σήμερα στην Ευρώπη να κάνουμε μια ενιαία αγορά στον ηλεκτρισμό και στην ενέργεια και από την άλλη εξακολουθούν ακόμα κράτη-μέλη και περιοχές της ε, Ευρώπης να είναι απομονωμένες από τα μεγάλα ηλεκτρικά ε, και ενεργειακά δίκτυα και εδώ ακριβώς έγκυται και ο ρόλος που μπορούν και διαδραματίζουν οι ρυθμιστικές αρχές ενέργειας σε ε, εθνικό επίπεδο. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς μπορεί να ε, βελτιώσει αυτή τη σχέση και τη συνεργασία ο Acer με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ώστε να μπορέσουν πρώτα πρώτα να, να περιοριστεί να αρχή αυτή η απομόνωση αλλά να βελτιωθεί και η τροφοδοσία ε, σε ενέργεια να υπάρξει δηλαδή ενεργειακή ασφάλεια και στα κράτη-μέλη, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ιδιαίτερα στη σημερινή κατάσταση χρειάζεται να υπάρχει ε, και μια εθνική ευελιξία και ανεξαρτησία για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους ε, σε ενέργεια αρκετά κρατημέλη. Και το ερώτημα που προκύψει ακριβώς είναι αυτό, πώς μπορεί να ενισχύσει ο ΕΣΕΡ την ε, συνεργασία σε αυτήν την κατεύθυνση με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you very much, Madam Werner. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βέρνερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι οι ανθρώπινοι πόροι δεν είναι απλώ λίγοι, αλλά θα μπορούν να εκπληρώσουν και τις υποχρεώσει. Έχουμε τις εθνικές εθνικές αρχές, θα μπορούσαμε να τι επιβαρύνουμε, ε, τι αποφορτήσουμε. Μήπω θα μπορούσατε να απορροφήσετε επομένω προσωπικό από τι εθνικέ ρυθμιστικέ αρχέ στο Racer. Ίσως ήταν αυτό μια δυνατότητα για να είστε ικανοί να επιτελέσετε το έργο σα και να υποστηρίξετε τα συμφέροντα. Well, thank you so much. I'm sorry. Ευχαριστώ πολύ. <coughs> Δεν άκουσα την παρουσίαση, αλλά έχω μια ερώτηση. Συγγνώμη, ρωτήσα κάτι που ήδη έχουμε αναφέρει. Είναι ένα θέμα που έχω θέξει και στο παρελθόν, που είναι η αιτήσια έκθεση παρακολούθησης και την δημιουργία ικανοτήτων διασυνοριακών, όχι μόνο φυσική ικανότητα, αλλά και διαθεσιμότητα διασυνοριακών ανταλλαγών και αυτό το θέμα έχει να κάνει με το αν έχουμε πρόσβαση σε αυτό το τομέα, σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να το δείτε αυτό το θέμα και να το ε, εντάξετε στην έκθεσή σας γιατί θα αποτελέσει πολύ χρήσιμο ε, εργαλείο για την ελεύθερη ροή πληροφοριών, τη διασυνοριακή ροή πληροφοριών. Σας στείλαμε μια επιστολή τον περασμένο Νοέμβριο για αυτό το θέμα και θα ήθελα να ξέρω αν το εξετάσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Τορσενόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Μίλησαμε πολλές φορές για την σημασία του οργανισμού Acer και για το πρόγραμμα REMIT και πάντα λέμε ότι έχουμε ανησυχίες ως προς την και θα τα καταφέρει, αν θα μπορέσει όλο αυτό το πακέτο των δεδομένων στο πλαίσιο του Ρέμιτ να τα επεξεργαστεί. και αν θα είναι δυνατόν να επεξέλθει στις ε, υποχρεώσεις. Πολύ σημαντικό ε, θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενέργεια και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συγκεκριμένους ε, κανονισμούς και διαδικασίες ε, αναβάλουμε τις πρωτοβουλίες μας. Από την Επιτροπή μας έχετε μία άτυπη υποστήριξη, η οποία είναι μέγιστη, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να περιγράψουμε αυτή την κατάσταση από κοινού με τη συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, γιατί από εκεί ξεκινάει να εξελίσσεται όλο το σύστημα. Δεν είμαι υποστηρικτή μιας ενιαίας ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής, φαντάζομαι ότι το κατανοείτε αυτό. Ίσως θα άξιζε, λοιπόν, να έχουμε μια μεγάλη έκθεση για τον οργανισμό Acer, να την επεξεργαστούμε και να αναφερθούμε και στη σημασία που έχει ο οργανισμός αυτός για την Ευρώπη. Μας ενημερώσατε για το βαθμό εφαρμογής του τρίτου ενεργειακού πακέτου σε γενικές γραμμές. Θα μπορούσατε να μας πείτε σε ποσοστά πόσο είναι το επίπεδο εφαρμογής, γιατί υπάρχει μια σάφια. Δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Πού βρισκόμαστε. Παραδείγματο χάρη, κωδική, ε, ποσοστά μετάδοση μεταξύ κρατών μελών. Ίσως ήταν επικίνδυνο να φέρουμε σε παραδείγματα συγκεκριμένων κρατών μελών. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά πάλι θα θέλαμε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία γιατί είναι δύσκολο ε, αλλιώς να παρεμβούμε στα κράτη-μέλη. Όπως είπαν κάποιοι συναδέλφοι θέλουμε να βοηθήσουμε, να σας βοηθήσουμε, αλλά δεν ξέρουμε την πραγματική διάσταση των πραγμάτων στα κράτη-μέλη. Και ένα δεύτερο θέμα έχει να κάνει με το λεγόμενο hardware στην εσωτερική ενεργειακή αγορά. Στην αγορά του φυσικού αερίου είναι η δυνατότητα να ε, χρησιμοποιούμε αντίστροφε ροέ. Γιατί να μην, ίσως δεν υπάρχουν αρκετέ διασυνδέσει, αλλά είναι αρκετέ. Σε ποσοστά λοιπόν, μπορείτε να μας αφαιρθείτε πόσα είναι τα ποσοστά των αντίστροφων ροών. Διαφορετική είναι η κατάσταση όμως στην ε, αγορά του ηλεκτρισμού. γιατί το επιθυμητό είναι το 10% της ε, χρήσης της ενέργειας στα κράτη-μέλη. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Είμαστε επίπεδο του 3%, 7%. Θα πετύχουμε το, έχουμε πετύχει το 10% σε κάθε κρατός μέλος. Έχει να κάνει με το hardware και με το software. Τα ποσοστά μετάδοση φυσικά είναι επίσης πολύ σημαντικό ε, οι ρυθμισμένες ε, τιμές επίσης, γιατί είπατε ότι θα τεθεί σε ισχύ η οδηγία για το REMIT Μεγάλο το όνομα της οδηγίας, κάνει μνήμα και στην δακαιρεότητα και στη διαφάνεια. Πώς είναι η ώρα να έχουμε ρυθμισμένες τιμές ε, σε κάποια κρατημέλη. Απίστευτες επίσης πρωτοβουλίες σε κάποια άλλα κράτη-μέλη, διαφορετικές πρωτοβουλίες ε, σε κράτη-μέλη για ε, ορυκτά καύσιμα, για πυρηνική ενέργεια, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λοιπόν, ε, προς τα πού βαδίσουμε στο να σταματήσουμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες μέχρι το 2020 θα ήταν υπέροχο να μπορούσαμε να πούμε ότι το 2020 θα σταματήσουν όλες αυτές οι πρωτοβουλίες. Έχουμε πολλά τέτοια ερωτήματα που αφορούν το hardware, το software, την, ε, το REMIT και παράλληλα δεν αναφέρατε ποια είναι η διαφορά στην περίπτωση της οδηγίας REMIT ε, ανάμεσα στο αέριο και στην ηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχει μεγάλη διαφορά κατά την άποψή μου. Ίσως ε, να μην ήμουν και αρκετά προσεκτικός ε, και να μην το πρόσεξα, αν το αναφέρατε ήδη, αλλά θα ήθελα πιο πολλές ε, πληροφορίες. Ε, δεν βλέπω κάποιον άλλο θέλει να θέσει ερωτήματα, οπότε ο λόγος και πάλι σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες ε, ερωτήσεις. Να ξεκινήσω με το θέμα των πόρων και του προϋπολογισμού, όπως επίσης και με την ε, ε, δυνατότητα υποστήριξής μας από τους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς, σε κάτι που έθεσε νομίζω η κυρία Κάλες, η κυρία Βικούνεν, νομίζω ο κύριος Σιλικιώτης επίσης το έθεσε. είναι θέμα προπολογισμού, αλλά είναι και θέμα εμπειρογνωμοσύνη. Αν δεν έχει κανεί ε, προπολογισμό για να προσλάβει του κατάλληλου ανθρώπου, τότε είναι μόνο θεωρητικό το θέμα τη εμπειρογνωμοσύνη. Πρέπει να πω ότι με του πόρου, με τον προπολογισμό που έχουμε στη διάθεσή μα, ήμασταν μάλλον τυχεροί. Καταφέραμε να ε, έχουμε κάποια αποτελέσματα ε, και να προσλάβουμε νέους αλλά ε, πολύ ε, ικανούς και αρκετά έμπειρους ε, ανθρώπους η ομάδα εποπτείας είναι μόνο τρία άτομα, αλλά πόσο μπορώ να κρίνω είναι πολύ καλή. Δεν μιλάμε για εκατοντάδες ανθρώπων, μιλάμε για ομάδες 10-20 ε, ατόμων που εξετάζουν την ε, αγορά, ε, όπως επίσης και τη συμπεριφορά των διαφόρων συμμετεχόντων στην αγορά. μπορεί να είμαστε τυχεροί δεν ξέρω πόσες φορές ε, η αντίστοιχη υπηρεσία στις Ηνωμένε Πολιτείε το υποδειγματική. Ήμασταν πραγματικά πολύ τυχεροί που μπορέσαμε να προσλάβουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορούσε να αντέξει την πίεση αλλά παρόλα αυτά ε, ήταν πάρα πολύ πεπειραμένος και εκπαίδευσε ολόκληρη την ομάδα. Δεν μιλάμε λοιπόν για τεράστιο αριθμό ατόμων, απλώς πρέπει να χρειαστεί, να, πρέπει να είμαστε τυχεροί μερικές φορές Δουλεύουμε πολύ με τους εθνικούς ρυθμιστικού φορείς. Νομίζω ότι την έδωσα αυτή την εντύπωση, ελπίζω τουλάχιστον. Ε, ο οργανισμός μας ε, παρακολουθεί την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά επίση παρακολουθεί και τις εθνικέ ε, αγορές με βασική αρμοδιότητα βέβαια. Αυτό είναι βασική αρμοδιότητα και ευθύνη των εθνικών ρυθμιστικών φορέων. Μερικές φορές έχουμε αναλάβει ε, νέα καθήκοντα και γι' αυτό έχουμε προσλάβει και επιπλέον προσωπικό. Πάντως οι πόροι μας είναι πολύ περιορισμένοι. Ε, επομένως το ίδιο καζάνι βράζουμε. Προσπαθήσαμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε ε, τη συνεργασία μας, αλλά με πολύ περιορισμένους πόρους και αυτό πραγματικά αποτελεί μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Μερικές φορές μάλιστα είναι και αδύνατο. Υπάρχει και υπήρξε ένα ερώτημα πώς οι εθνικές ε, ρυθμιστικές αρχές και οργανισμός μας ε, μπορούν να απομακρύνουν ε, τις ενεργειακές νήσους. Κοίταξε τι να σας πω. Είναι θέμα υποδομής εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Έχουμε προσπαθήσει να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα με νομοθεσία που πέρασε το 2013. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε την υποδομή σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μην υπάρχουν αυτοί. Ε, αυτές οι ε, ε, ο Acer και οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές ε, εργάζονται πολύ ε, σκληρά για τις επιλογές των απαραίτητων προγραμμάτων και τη παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών, όπως επίσης και τον εντοπισμό οποιονδήποτε εμποδίων μπορούν να καθυστερήσουν την εξέλιξη. Αναφέρθηκε επίσης η επιστολή πολλών ευρωβουλευτών σε σχέση με τις διασυνοριακές ε, ε, συναλλαγές. Είναι κάτι το οποίο θα το ε, επεξεργαστούμε αυτή τη χρονιά, προσπαθούμε να συλλέξουμε δεδομένα, έχουμε καταφέρει να ε, συλλέξουμε κάποιες πληροφορίες. Νομίζω ότι περιμένουμε την ε, έκθεση τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου και ελπίζω να μπορέσω να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα και να, να δούμε κατά πόσο η ανάλυση που κάναμε εμείς ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας. Για μας πάντως αυτό αποτελεί προτεραιότητα. Τώρα πώς εσείς ως Επιτροπή και το ε, Κοινοβούλιο στο σύνολό του ε, μπορείτε να βοηθήσετε. Έχουμε συνεχή σχέση, συνεχείς επαφές με την ομάδα, μέσω της ομάδας επαφών και έχουμε ε, θέσει στη διάθεσή σας κάποια ενημερωτικά σημειώματα που εξηγούν τη δική μας δουλειά και τη δουλειά του Remit και αφορά τις προκλήσεις, ε, την ε, εργασία μας, ε, μία μη απόρριτη σύνοψη των διαφόρων υποθέσεων που διαχειριστήκαμε από κοινού με τις εθνικές αρχές και υπάρχει επίσης και μία βαθμολόγηση των ε, δραστηριοτήτων μας. Ε, αν μου το επιτρέπει ο Πρόεδρος, εγώ ευχαρίστως να σας διανύμω τη συγκεκριμένη έκθεση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ανάγνωσμα. Το δικό σας ερώτημα. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω αλλά δεν ε, θυμάμαι όλους τους, ε, όλα τα νούμερα αυτή τη στιγμή. Η εφαρμογή του ενεργειακού κεκτημένου στα κράτη-μέλη, που είναι, είναι κάτι το οποίο το παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμείς εφαρμόζουμε το τρίτο πακέτο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορώ να σας δώσω κάποια στατιστικά στοιχεία. Ε, όταν ε, μιλάμε για παράδειγμα για τους κανόνες, οι τρεις από τις τέσσερις, οι τρεις, από τους τέσσερις κώδικες δικτύου για το αέριο έχουν εγκριθεί. Νομίζω ότι υπάρχει ένας ο οποίος είναι σε κρεμότητα στον ηλεκτρισμό, ένας έχει περάσει και θα αρχίσει να ισχύει μέχρι το τέλος της χρονιάς και οι υπόλοιποι ε, βάσει του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα περάσουν από την Επιτροπολογία αυτή τη χρονιά εκτός από ορισμένους που συνδέονται με την πρωτοβουλία που αφορά τις ενεργειακές αγορές. Ε, για τις ρυθμιζόμενες τιμές, δύο τρίτα των χωρών εξακολουθούν να έχουν τέτοιου είδους τιμές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, όχι μόνο όταν είναι χαμηλότερες του κόστους, ε, αυτό είναι ένα απόλυτο εμπόδιο, αλλά και μερικές φορές και όταν είναι πάνω όταν είναι ε, πάνω από το κόστος. Τώρα, ε, η διασύνδεση, ε, το επίπεδο διασύνδεσης σε μερικές περιπτώσεις ε, έχουμε πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα στην ε, Ιβρική Κερσόνησο έχουμε ένα 10% απόκληση από τον υπόλοιπο μέσο όρο σε μεγαλύτερο βαθμό, σε γενικές γραμμές όμως υπάρχει ένα αρκετά καλό επίπεδο διασύνδεσης σε μερικές περιπτώσεις ε, δεν έχει γίνει άλλωστε διασύνδεση των διαφόρων αγορών και μερικές φορές οι ροές πηγαίνουν προς λάθος κατεύθυνση και αυτό είναι κάτι που καταστρέφει ε, την ε, αξία για τους καταναλωτές. Είναι σαν να πετάμε λεφτά από το παράθυρο. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές στην Ευρώπη δεν θα πληρώνουν παραπάνω από αυτό που είναι απολύτως απαραίτητο για τις αντίστροφες ροές. Νομίζω ότι στα περισσότερα σύνορα εφαρμόζεται πλέον το σύστημα των αντίστροφων ροών. Μάλιστα, δεν πολύ άσχημα, λέει ο Πρόεδρος. Έχετε το λόγο. Ναι, θα ήθελα... Το θέμα των, της συνεργασίας ανάμεσα στις ρυθμιστικές αρχές και το Acer. Εμείς έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο ύπαρξης. Νομίζω ότι αυτό το οποίο αποδείξαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι μπορούμε να βοηθήσουμε στη στενή συνεργασία μέσω της επικοινωνίας. Έχει υπάρξει υποστήριξη κάτω από οικονομικές συνθήκες σχετικά περιορισμένες και κάτω από συνθήκες λειτουργίας των ρυθμιστικών αρχών επίσης ε, ε, περιορισμένες. γίνονται αποσπάσεις στις υπηρεσίες μας για ένα-δύο χρόνια ή και για μικρότερη χρονική διάρκεια από πλευράς των ρυθμιστικών αρχών. Οι υπηρεσίες του Συμβουλίου μας παρέχουν άλλες ε, ε, διευκολύνσεις για πολλές από τις συναντήσεις που γίνονται εδώ ε, στις Βρυξέλλες. Υπάρχει σε αιτήσια βάση επιμελητιακή στήριξη που ξεπερνά πάνω τις 100.000 από πλευράς των ρυθμιστικών εθνικών αρχών. Και για το ρήμιτ υπάρχει ενίσχυση και βοήθεια στα πλαίσια των ομάδων εργασίας. Δηλαδή, να σας το πω με λίγα λόγια, υπάρχει στενή συνεργασία ανάμεσα στις ρυθμιστικές αρχές. Τώρα, για το αν μπορούμε να μιλήσουμε για ενιαίο σύστημα. Ε, αυτό είναι πολύ πολιτικό θέμα κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων αυτή που εγώ γνωρίζω καλύτερα, δεν θα ήθελα να υπάρχει μια κεντρική ρυθμιστική αρχή. Υπάρχουν πάντως σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις εθνικές αγορές και η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς θα τις καταργήσει και τότε σε πολιτικό επίπεδο τα πράγματα θα γίνουν πιο απλά. Δεν θέλω να μπω βαθύτερα στην πολιτική διάσταση, αλλά νομίζω ότι έχουμε την δυνατότητα με τους μειωμένους πόρους ε, να συνεργαστούμε ακόμα πιο στενά. Thank Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για όλες τις παρατηρήσεις σας και τις εξηγήσεις σας. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα η εσωτερική αγορά και γι' αυτό θα θέλαμε πριν το τέλος του χρόνου να σας ξανασυναντήσουμε και να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες και στατιστικές. Ελπίζω οι στατιστικές, τα στατιστικά στοιχεία τότε να έχουν βελτιωθεί πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και τις εξηγήσεις σας. Well, dear colleagues, ladies and gentlemen, unusual guests, unusual guests. Συνήθις του φιλοξενούμενοι. Ήσαν ο Γενικός Διευθυντής και ο Πρόεδρος του Acer. Ήταν αναμενόμενοι επισκέπτες, αλλά στην περίπτωση τώρα του σημείου 13 της ημερήσιας διάταξης ορίζον 2020 θα συζητήσουμε με τον Ζαν Πιερ Μπουργκινιό, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και δύο νέους επιστήμονες, δύο νέους επιστήμονες Χαίρομαι που σας συναντώ και τους δύο. Συναντηθήκαμε πριν λίγες ώρες με τον κύριο Μπουργενιό. Να σας υπενθυμίσω συναδέλφοι ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ερευνάς δημιουργήθηκε στα πλαίσια του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη και νιώθω υπεύθυνο γι' αυτό γιατί ήμουν εισηγητής για το 7ο πρόγραμμα. Έχει ε, τύχει πλήρους ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αναγνώρισης το Συμβούλιο αυτό. Χάρη στο Συμβούλιο αυτό νομίζω ότι μπορέσαμε να κρατήσουμε τους νέους επιστήμονες στην Ευρώπη και μπορέσαμε επίσης να προσελκύσουμε στην Ευρώπη και άλλους ερευνητές. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω από τον καθηγητή αν κάτι τέτοιο ισχύει και αν μπορεί κανείς να ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι το Συμβούλιο σε κάποια φάση αποφάσισε να διπλασιάσει ε, τις πιστώσεις ε, σε σχέση με τα 6,5 εκατομμύρια τα οποία είχε δώσει στο παρελθόν. Η Επιτροπή Ήτρε λοιπόν και η κυρία Βαν Μπρέμπτ επιτυχώς αντιστάθηκε θα έλεγα στις επιθέσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ήταν ένα από τα τρία θέματα τα οποία δεν υπέστησαν μειώσεις. Είναι μεγάλο επίτευγμα λοιπόν το ότι μπορούμε να υπερασπιστούμε τον προϋπολογισμό αυτό. Και η Επιτροπή ε, προσπαθεί τώρα ή μάλλον παρακολουθεί καλύτερα τις εργασίες αυτού του Συμβουλίου όπως και εμείς που κάναμε αυτή την τεράστια προσπάθεια ε, να ε, σας υπερασπιστούμε, περιμένουμε πολλά, κάνατε ήδη πολλά Θα κάνετε την εισαγωγική σας παρατήρηση και μετά η κυρία Τόλιτς από την Κροατία και ο κύριος Πούνιο από την Ιταλία θα παρουσιάσουν τις δικές τους απόψεις για το πόσο βλέπουν το Συμβούλιο αυτό και την δυνατότητα συνεργασίας επί τη βάση του προγράμματος. Έχετε να μας παρουσιάσετε τις προσωπικές σας εμπειρίες, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να πάρω το λόγο. Την ημέρα που το Ευρωπαϊκό ε, Συμβούλιο Έρευνας υπογράφει το ε, το, ε, συμβόλε το πολλωστό του συμβόλαιο, ε, ε, η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, ειδικότερα η δική σας επιτροπή έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ε, δεχθήκατε επίσης να είναι εδώ ο Νικολά ε, Πουνιό, ο οποίος μπορεί να μας πει ορισμένα πράγματα στο πλαίσιο της σύμβασής του με το Συμβούλιο Έρευνας και η κυρία Τόλιτς, η οποία θα μας πει για το πώς η συμμετοχή της στο Συμβούλιο Έρευνας εντάσσεται στην επιστημονική της καριέρα. 7-8 ε, χρόνια ε, πριν αρχίσαμε την προσπάθεια αυτή. Το 2009 ε, αρχίσαμε να αποτελούμε ένα σημαντικό παίκτη στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έρευνας. Τι έχουμε κάνει εδώ και 8 χρόνια πάνω από 15% των ε, αξιολογητών ε, της Ευρώπης προέρχονται εκτός, από, από, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να πούμε ότι ε, σε κάθε διαγωνισμό 600 επιστήμονες έρχονται για να κάνουν την επιλογή και μιλάω για 95 διαφορετικές εθνικότητες. 9 δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση πάνω από 5 εκατομμύρια ε, προγραμμάτων ε, σε 32 χώρες ε, της Ευρώπης από 166 εθνικότητες, 40.000 ερευνητές, 9.000 διδακτορικούς και 4.000 ε, μεταδικτατορικούς. Ε, το 2016 θα γίνει μια ε, έκθεση που θα αξιολογήσει πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας για όσους έχουν μια μετέπειτα επιστημονική καριέρα. 48 άρθρα ε, έχουν αναφερθεί στο θέμα αυτό σε επιστημονικές επιθεωρήσεις και υπάρχουν επίσης και ε, πολλές επιθεωρήσεις ε, που αναφέρονται συγκεκριμένα στους στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας ώστε η έρευνα να, είναι, να έχει μια καλύτερη θέση στο πλαίσιο των επιστημονικών επιθεωρήσεων. Ε, πέντε βραβείο Νόμπελ ε, είναι, ε, ένα από τα, είναι μια πολύ σημαντική ένδειξη της σημασίας του Συμβουλίου Έρευνας Είμαστε πραγματικά, είναι πραγματικά μια πολύ ωραία περιπέτεια. Εγώ γνωρίζω ε, το, ε, την Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας από τις απαρχές του, ε, όταν υπήρχε ο, ο απλός οργανισμός επιστημονικής κοινότητας και μετά εδώ και 1,5 χρόνο είμαι πρόεδρος της, του νέου Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Ε, είναι πραγματικά ένα μοναδικό, ε, μια μοναδική προσπάθεια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, είναι υπεύθυνο και για την οργάνωση της εκτίμησης των διαφόρων προγραμμάτων. Δεν, δεν, δεν, δεν αναφέρεται η προτεραιότητα. Οι βάσεις οι αρχές βάσεις, ε, δηλαδή ε, κρίση βάση της επιστημονική ποιότητας των προγραμμάτων, ε, μεταξύ άλλων, έχουν καταδείξει τη σημασία τους σε επιστημονικό επίπεδο. Είναι ευέλικτη η χρηματοδότηση, μακροπρόθεσμη για πέντε χρόνια, σε επιστήμονες που παρουσιάζουν φιλόδοξα προγράμματα για να μπορέσουν να παρουσιάσουν τις εργασίες τους στην Ευρώπη. Και μία φορά ακόμη γίνεται ε, ανεξαρτήτως προτεραιότητας των επιστημονικών τομέων. Είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός 10% είναι το ποσοστό ε, επιτυχίας. Ε, έχει αναγνωριστεί η μέθοδος αυτή ένας από τους καλύτερους τρόπους ε, για να μπορέσει κανείς να προβεί σε επιστημονικές επαναστατικές ανακαλύψεις. Μέχρι τώρα δύο τρίτα της χρηματοδότησης έχουν αφιερωθεί σε νέους ερευνητές, κάτι που θα συνεχίσει. Μέχρι το 2012 ο προϋπολογισμός ε, τα τρία πρώτα χρόνια 100 εκατομμύρια λιγότερα από ε, το 2010 ε, έγινε όμως μια μεγάλη αύξηση, έχουμε φτάσει τα 13 δισεκατομμύρια. Η επόμενη αύξηση ε, θα γίνει το 2018 μέχρι το 2020. Ε, αυτή τη στιγμή βέβαια το 10% ποσοστό επιτυχίας θα παραμείνει εκτός αν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές για, στις πιστώσεις τις διαθέσιμες. Η κατάσταση αυτή είναι απογοητευτική γιατί μας δημιουργεί προβλήματα στις νέες προτάσεις που θέλουμε να κάνουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να αρνηθούμε ορισμένα εξαιρετικά ε, προγράμματα σε ζητήματα μηχανικής για παράδειγμα ή πιο τεχνικά ε, προγράμματα. Πρέπει να προοδεύσουμε ε, την ε, έρευνα μεταξύ των διαφέρων επιστημονικών τομέων, ε, στην οποία συμμετέχουν πολλοί νέοι επιστήμονες. Ε, έχουμε ζητήσει να υπάρξουν εταιρικέ σχέσεις μέσω διαγωνισμών 2012-2013. Δυστυχώς όμως δεν υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συνεπώς ε, πολλές ε, κοινότητες υποεκπροσωπούνται, οι γυναίκες για παράδειγμα, ειδικότερα στο τομέα ε, που, σε τομείς που είναι πολύ σημαντικοί για την Ένωση, ερευνητές από χώρες που το ποσοστό επιτυχία τους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας είναι χαμηλότερο. Ε, το επίπεδο αυτή τη στιγμή ε, του προσωπικού και των διοικητικών ε, εξόδων ορίζεται για 7 έτη. Μπορώ να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα ε, για κάποια καμψία που υπάρχει. Για παράδειγμα, χρειάζεται ο ίδιος διοικητικός χρόνος για να υπάρξει ένα, μια σύμβαση για μικρότερο ή μεγαλύτερο πρόγραμμα. Ε, δηλαδή, την ίδιο χρόνο θα κάνουμε για να υπάρξουν κάποιες διερευνητικές εργασίες, για παράδειγμα, ε, όπως θα χρειαστεί για ένα μεγαλύτερης κλίμακας πρόγραμμα. Όπως γνωρίζετε, το, στα τέλη του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει μία αναθεώρηση της κατάστασης έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θα θέλαμε να συμμετέχουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν να δείξουν ότι υπάρχουν νέες προτεραιότητες. Πολύ συχνά ε, χρειάζεται να ε, η υπάρξει καινοτομία, πρέπει να επαγρυπνούμε, πρέπει να αντιδρούμε στις προκλήσεις, πρέπει να έχουμε ε, ε πρωτοβουλίες. Ε, δεν είναι μόνο θέμα χρηματοδότησης. κάθε φορά που τίθεται ένα σημαντικό, πρόγραμμα, ένα σημαντικό πρόβλημα πρέπει να χρηματοδοτούνται οι έρευνες εκ των προτέρων. Το Global Research Council ε, θα συνεδριάσει φέτος στο Τόκιο. η υπεύθυνη χρηματοδότηση των ερευνητικών Ινστιτούτων ε, τεράστιας ε, παγκόσμιας σημασίας θα συμμετέχουν. Το να μπορέσει να γίνει όμως κάτι τέτοιο τόσο σύντομα μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω τη βοήθειά σας. Πρέπει να υπάρξουν ε, ε, να υπάρξει συνεργασία με ε, τη National Research Foundation των Ηνωμένων Πολιτειών, με ερευνητικά Ινστιτούτα της Αργεντινής. Έχουν υπάρξει τέτοιου είδου συμφωνίε το 2015. Υπάρξει μια τέτοια συμφωνία που έχει δρομολογηθεί με την Κίνα και με την Ιαπωνία. Αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι η αναγνώριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας σε παγκόσμιο επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Uh, Η κυρία Τόλιτς έχει το λόγο. Έχετε το λόγο. Ε, Ονομαμαι Βατόλη, έχω λάβει υποτροφία φέτος για να σπουδάσω βιοφυσική στο Ρούσερ Μπός της Ινστιτούτου του Ζάγκρεμπ. Να σας μιλήσω πρώτα για την καριέρα μου. Κατάγομαι από το Ζάγκρεμπ, όπου σπούδασα μοριακή βιολογία. Έκανα τεκτονική μου διατριβή, αλλά κατά τη διάρκεια της αρχιτεκτονικής μου διατριβής κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να ασχολήθηκα με την επιστήμη πως θα ήθελα και γι' αυτό πήγα στην ε, Βοστόνη που ολοκλήρωσα το PhD μου στο Harvard. Έκανα αίτηση για μεταδεκτορικά το ένα στην Κοπεχάγη και το άλλο στην Φλωρεντία. Και μετά από αυτέ τι εκπαιδεύσει έγινα ε, ερευνήτρια στο Glang Institute στην Δρέσδη όπου πέρασα 10 χρόνια ε, κάνοντας έρευνα σε ένα εκπληκτικό περιβάλλον. Μετά από αυτή την ε, ε, εκτεταμένη εμπειρία που απέκτησα, αποφάσισα να επιστρέψω στην γενέτειρά μου το Ζάγκρεμπ. Πήγα λοιπόν στο Ρούζερ Μπόσκεβιτς Ινστιτούτο, έγινα καθηγήτρια, προτού να λάβω την υποτροφία στο ERC. γιατί ήθελα να ασχοληθώ με την έρευνα στο επίπεδο που τα έκανα και στο Max Planck στη Γερμανία, όμως ε, είχα ανησυχίε για την ε, χρηματοδότηση και όπως καταλαβαίνετε οι επιτροφές που χωρούνται από το κροάτικο κράτος είναι πολύ πενιχρές. Το ERC μου έδωσε την απάντηση και χάρη στην υποτροφία ε, μου δόθηκε ευκαιρία να δημιουργήσω μια ομάδα ερευνητών ε, τρεις μεταδιδακτορικούς ε, φοιτητές, δύο μεταδιδακτορικούς ε, φοιτητές και ε, τους προσέλαβα και κατάφερα να αγοράσω τον εξοπλισμό και τον μικροσκόπιο που χρειαζόμασταν για την έρευνά μας και για τα πειράματά μας. Τα πειράματά μας ε, έχουν να κάνουν με, την, με τους με τη διάσπαση ε, και πρόκειται για μια διαδικασία που δεν ξέραμε ακριβώ πώ λειτουργεί. Στο πρόγραμμα μα προσπαθήσαμε να βάλουμε σε εφαρμογή ε, όλε τι γνώσει που είχαμε στη διάθεσή μα. Και το βασικό ερώτημα είναι πώς ε, το κέλυφος διαχωρίζει τα χρωμοσώματα σε δύο κομμάτια χωρίς να υπάρξουν λάθη. Υπάρχουν ε, μικρή, μικρά στέλεχη από πρωτεΐνες που ε, ε, προσκολώνται στα χρωμοσώματα. Και φυσικά αποτελούν και στόχο των ε, χημιοθεραπείων γιατί κατά αυτόν τον τρόπο αποτρέπουν την διάδραση ανάμεσα στα χρωμοσώματα και αποτρέπουν φυσικά την εξέλιξη του καρκίνου. Αυτά ε, κινούν τα χρωμοσώματα μπροστά και πίσω και στη συνέχεια τα διαχωρίζουν. Στη συνέχεια τα χρωμοσώματα πηγαίνουν στην άλλη άκρη του κυτάρου και ξέρουμε ότι τα microtubules έχουν, ε, ε, διαδρούν ε, με τα χρωμοσώματα αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι οι παράμετρες της διάδρασης. Μόνο τα microtubules που ε, έχουν διάδραση με τα χρώσματα στις άκρες τους μπορούν ε, να έχουν αυτή την ε, διάδραση. Υπάρχουν βέβαια και άλλα τέτοια ευρήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν διερευνηθεί παρκώς με τη χρήση των πιο εξελιγμένων μικροσκοπίων και οργάνων μπορούμε να ορίσουμε τις πρωτεΐνες που ε, τα συνδέουν αυτά και αυτές οι πρωτεΐνες συνέχεια μπορούν ε, να αποτελέσουν ε, κομμάτι της θεραπείας κατά του καρκίνου. Έχουμε μία διατομιακή προσέγγιση, έχουμε την μοριακή βιολογία, γενετική, μικροχειρουργική, πληροφορική και φυσική για να ε, διερευνήσουμε, για να ερευνήσουμε αυτό τον κλάδο. Και ενδεχομένως... Ε, the mitotic anti-cancer strategies because microtubules are a major target ε, for chemotherapy. Ε, και οι μικροσωλήνες είναι πολύ σημαντικοί γιατί αποτελούν βασικό στόχο την χημειοθεραπεία, στην βιοιατρική, η βασική έρευνα στη βιολογία είναι το κλειδί που ανοίγει νέους δρόμους για την εφαρμογή ε, μεθόδων, ώστε να βρούμε τρόπους, ε, νέους τρόπους θεραπείας και διάγνωσης ε, πλήθους ε, παθήσεων και ασθενειών. Ο καθοριστικός ρόλος του ERC χρηματοδοτώντας την βασική έρευνα που μακροπρόθεσμα θα έχει αντίκτυπο στην κοινωνία. Ευχαριστώ κυρία. Τόλιτς. If I may to ask our uh, second young scientist, Mr. Πούνιο. Στον κύριο Πούνιο. Ο λόγος στον κύριο Πούνιο. Grazie molte, eh, signore e signore. Eh, un, un... Ε, Είναι τιμή μου και ευχαρίστηση που βρίσκομαι εδώ σήμερα μπροστά σας. Θα ήθελα να παρουσιάσω τη δική μου προσωπική εμπειρία και την ερευνητική μου δραστηριότητα που χρηματοδοτήθηκε από το Συμβούλιο Έρευνας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Εγώ προσθέτω εδώ την προσωπική μου εμπειρία που ξεκινά το 2010 όταν αποφάσισα να ζητήσω μια υποτροφία, τότε δεν ήξερα ακριβώς πώς χρηματοδοτεί ε, το European Research Council. Αποτέλεσμα ήταν ότι η πρότασή μου δεν έγινε δεκτή γιατί τα στοιχεία τα οποία είχα δώσει δεν ήταν ικανοποιητικά. Εγώ εξεπλάγιν βέβαια από τον ε, υψηλό αριθμό των ελεγκτών αναθεωρητών οι οποίοι είπαν ότι το κουρίκουλουμ βίτε μου ήταν ισχυρό αλλά η έρευνά μου δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένη. Χρειάστηκε λοιπόν να υποβάλουμε εκ νέου τον επόμενο χρόνο την πρόταση έρευνας αρκετά ενδυναμωμένη θα έλεγα και μπορέσαμε να παρουσιάσουμε λοιπόν την πρόταση αυτή με προφορικό τρόπο σε επίπεδο συνέντευξης δηλαδή εδώ στις Βρυξέλλες έγινε η παρουσίαση και πήρα την υποτροφία. Χάρη στην υποτροφία αυτή το Πανεπιστήμιο του Τρέντο, το οποίο είναι ιδιαίτερο στην Ιταλία, αλλά ασχολείται πάρα πολύ με τα θέματα αυτά, έχει θα έλεγα πάρα πολλούς υποτρόφους του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού, και εγώ ε, δίδαξα στην αρχή σαν υφηγητής και μετά σαν τακτικός καθηγητής μετά από ένα χρόνο θα έλεγα κάποιων ε, δισταγμών αποφάσισα με τη γυναίκα μου και τα παιδιά να μετακομίσουμε όλοι στο Τρέντο και ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια σε αυτό το πανεπιστήμιο στο οποίο βρήκα μια επικοδομητική ατμόσφαιρα. Το πρώτο πράγμα το οποίο έκανα ήταν να αποκτήσω ε, ένα, ε, μια μηχανή έρευνας, δοκιμαστική μηχανή με μικροσκόπια, νανοσκόπια που ελέγχει σε επίπεδο μηχανικής αντοχής τα υλικά ε, μπορέσαμε να έχουμε και κάποιες υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές και για μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Στήσαμε λοιπόν ένα μικρό θα έλεγα νανομηχανικής, ενεργαστήριο, εργαστήριο ακριβώς νανομηχανικής. Συνεργαζόμαστε με βιομηχανίες μεγάλες στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο και μπορούμε να δημοσιεύουμε πάρα πολλές εργασίες σε μηνιαία βάση. Η πρώτη εργασία την οποία κάναμε και ήμασταν τυχεροί γι' αυτό ε, πήρε το εξώφυλλο του περιοδικού Nature. Λοιπόν, ιεραρχικά υπερνανοηλικά λέγεται η η πρώτη εργασία και προσπαθούμε εμείς να βγάλουμε κάποια χαρακτηριστικά ανώτερα σε μηχανικό επίπεδο από τα διαθέσιμα υλικά. Αυτό μας έστρεψε κατά κάποιο τρόπο να πάρουμε και ένα δεύτερο πτυχίο στη φυσική και ένα δεύτερο διδακτορικό ε, το οποίο πήρα για να πω ότι εγώ ήμουν ε, θεωρητικός κατά κάποιο τρόπο μέχρι πριν λίγο καιρό. Μελετάμε λοιπόν πάρα πολύ ιδιαίτερα υλικά, να σας δώσω ένα παράδειγμα, δεν θα δώσω λεπτομέρειες. Ε, μιλάμε για το γραφήνιο σαν παράδειγμα, ε, το οποίο προέρχεται από τον άνθρακα αλλά είναι πολύ πιο ισχυρό από τον χάλιβα 100 φορές και άλλα υλικά επίσης, άλλες χημικές ουσίες οι οποίες ε, ε, είναι ισχυρότατες και κάποια χημικά στοιχεία. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν ε, από τα υλικά αυτά τα ειδικά τους χαρακτηριστικά υψηλής αντοχής. E anche per esempio la, la zampa del geco Έχουμε και άλλα παραδείγματα τα οποία μπορούμε να δώσουμε. Αναζητήσαμε και βρήκαμε κάποιους μηχανισμούς, βρήκαμε κάποιες ίνες ισχυρότερες κατά δέκα φορά, φορές από το κεβλάρ και έχουμε την δυνατότητα για βασική έρευνα για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου αυτού υλικού και για την δημιουργία επιφανειών οι οποίες είναι δυνατόν να είναι αυτοκαθαριζόμενες. Ε, ξέρετε τα υλικά που χρησιμοποιούμε όπως το χαλκό, όπως τον σίδηρο, την πέτρα. Η εισαγωγή ενός καταστροφικού οργανισμού μερικές φορές μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα του ανθρώπου. Αυτό είναι ο στόχος της επιστήμης και της τεχνολογίας και εγώ έχω ξεχάσει πολλές φορές να φάω για να επιδιώξω τον στόχο αυτό, αλλά μπορούμε νομίζω να πετύχουμε πολλά. Χωρίς όμως την βοήθειά σας και χωρίς τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Ταμείου δεν θα είχα κάνει τίποτα. Thank you. Thank Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. For our speakers from the hall, colleague Eller as a rapporteur Horizon 2020. Ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας στο θέμα αυτό. Χωρίς μικρόφωνο ο μιλητής. Εξακολουθεί ο μιλητής ε, να είναι χωρίς μικρόφωνο, δυστυχώς έχουμε υποχρεωτικά διακόψει. one Αυτό το μικρόφωνο πράγματι δουλεύει. Ευχαριστώ. Να σας ε, καλωσορίσω στο Κοινοβούλιο, κύριε Μπουργκινιόν. Είναι μια πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή ήταν πιο συγκρατημένη όσον αφορά την κατανομή του προπολογισμού. Υπάρχουν όμως κάποια θέματα που αφορούν τη χρηματοδότηση και θα προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε το ERC από τις ε, περικοπές. Θα ήθελα να σας κάνω ε, που αφορούν το μέλλον. Πώς βλέπετε την κατάσταση της έρευνας στην Ευρώπη. Έχουμε τις περικοπές το ERC ήταν επιτυχημένο ως προς ε, την άσκηση πίσω προς το lobbying, όμως έχουμε τεράστιες περικοπές. Και όταν βλέπω την κυρία Τόλιτς και το Ινστιτούτο στο Ζάγκρεπ, στο οποίο εργάζεται, και τη συνεργασία που θα μπορούσε να έχει με τη βιομηχανία, αυτό θα σημαίνει ότι θα υπήρξε πολύ μεγάλη, ε, ότι ενδεχομένω θα υπήρχαν ε, περικοπές στα πρόγραμματα έρευνα σε χώρε όπω είναι η Κροατία. 2,2 εκατομμύρια. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από το ERC, να έχουμε ξέχοντες επιστήμονες όπως εσάς και μετά να διευρύνουμε τη συνεργασία μας και τη δημιουργία δομών ε, σε τα νέα κρατημέλη, όμως εκεί λείπουν τα κονδύλια. Υπάρχει έλλειψη κονδυλίων. Ε, παρακαλώ την ΕΡΣΥ να προθίσει λοιπόν την έννοια της ελεγγύης και ε, με... Ε, ζητήσουμε στην επόμενη περίοδο του περιπολογισμού να ζητήσουμε από το ERC γιατί ε, δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας ε, ε, σε σχέση με άλλες χώρες όπως είναι η Νότια Κορέα κτλ. Δύο ερώτημα. Ένα, πώς βλέπετε την σύνδεση ανάμεσα στο ERC και την εξέχουσα δουλειά που παρουσιάζει και την διεύνηση της συνεργασίας στο ερευνητικό πεδίο και από την άλλη, μια ερώτηση στην αδελφό στην κυρία Τόλιτς. Πώς είναι η κατάσταση στην Κροατία. Προφανώς τώρα α, με την ε, υποτροφία του ΕΡΣΥ να μπορείτε να τα καταφέρετε, αλλά πώ θα, πώς θα συνεχίσετε στο μέλλον. Κυρία Μούντι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Είναι πολύ καλό να βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτών τα οποία συζητάμε στην Επιτροπή. Ειδικά με την προστασία που μπορούσαμε να έχουμε με τις ε, διαπραγματεύσεις σχετικά με το ERC, γιατί αυτή οι διάλογοι καταδεικνύουν την ε, σημασία των διατομιακών ε, θεμάτων που αφορούν όλες τις επιτροπές και τις ομάδες για τη χρηματοδότηση βασικής έρευνας. Να αναφερθώ σε δύο σημεία. Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό ήταν τόσο σαφής η προστασία Δεν είναι όπως μόνο το ERC που λαμβάνει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ορίζοντα 2020. Γιατί υπάρχει χρηματοδότηση και σε άλλα προγράμματα. Θα ήθελα λίγο να δείτε αυτό το θέμα και προφανώς ε, κατάγεστε από τον Ηνωμένο Βασίλειο και έχω προσωπικό συμφέρον στο να έχουμε θετική άποψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αφορά το μέλλον, πολλά από αυτά τα οποία συζητάμε και η χρηματοδότηση της βασικής έρευνας που είναι τόσο σημαντική για τη διασφάλιση του μέλλοντος που θέλουμε να έχουμε, ότι δεν πρέπει να επενδύουμε μόνο στην έρευνα της αγοράς, αλλά πρέπει να κάνουμε και ε, έγκαιρη έρευνα, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να είμαστε μπροστά στις εξελίξεις ε, στο μέλλον, στα, όχι στα επόμενα χρόνια, αλλά μακροπρόθεσμα. Θα ήθελα λοιπόν την άποψή σας από αυτού του θέματος. Μας είπατε τις ιστορίες σας, ε, τι μπορέσετε να πετύχετε μέσα από την έρευνά σας και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα παραδείγματα για να δώσουμε έμφαση στην προστιθέμενη αξία που έχει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στο ε, μέλλον μας. Ε, Ευχαριστώ, κυρία Κουντρίτσκα. Να συγχαρώ Ε, για τις υποτροφίες που έχουν χορηγηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Δεν είναι μεγάλη επιτυχία μόνο για το ERC αλλά και για τους ερευνητές που μπορούν να ολοκληρώσουν τα ερευνητικά τους προγράμματα. Δυστυχώς ανάμεσα στα επιτυχή προγράμματα δεν υπάρχουν τόσα πολλά από τα νέα κράτη-μέλη. Στο ERC υπάρχει μια ομάδα που ονομάζεται Επιστημονικό Συμβούλιο για την διεύρυνση της συμμετοχής που έχει ως στόχο να αυξήσει την συμμετοχή κρατών, ε, ερευνητών από λιγότερο ε, δραστήρια στην έρευνα περιοχές. Ποιοι είναι οι στόχοι αυτής της ομάδας, ποιες είναι οι της πρακτικές. Όταν αναλαμβάνει δράση το ΕΡΣΥ για να διασφαλίσει την καλύτερη ε, συμμετοχή. Δεύτερο σημείο η εγγραφή στο 5,5 ήταν το ποσοστό ε, συμμετοχή στον προπολογισμό του 7ου πακέτου. Ένα υψηλότερο ποσοστό ε, ε, μπορεί να μας... Ε, μπορεί στο μέλλον να μην έχουν ευκαιρίες για χρηματοδότηση κάποια μεγάλα project. Τι θα κάνει το ERC για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα και αν ε, είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση. Επόμενο ερώτημα. Όπως οι συνάδελφοι, χαίρομαι και εγώ για την παρουσία σας. Ξεκινάει το ε, υπαριθμό 5.000 πρόγραμμα είναι φυσικά πολύ δύσκολο το έργο σας, αλλά δείχνετε ότι υπάρχει πρόοδος και η, η παρουσίασή σας έγινε με συγκεκριμένα άτομα, με ερευνητές και αυτό αποτελεί κίνητρο για εμάς, για να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Και με ενδιαφέρει πολύ το θέμα που έθιξε ο κύριος Μπουρινιό. Ποιο θα μπορούσε να είναι το επόμενο βήμα ποια είναι η επόμενη αποστολή που θα πρέπει να ε, έχετε. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι το οικονομικό το κομμάτι θα αποτελέσει τόσο μεγάλο εμπόδιο. Πού θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες, σε ποιον τομέα. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βρικούνεν. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ ε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ε, ομιλητές, ε, τους προσκεκλημένους μας. Είναι πάρα πολύ καλό πάντοτε να έρχονται ερευνητές στην Επιτροπή μας γιατί η εκπαίδευση και η έρευνα, όπως γνωρίζουμε, είναι το κλειδί για το μέλλον της Ευρώπης και είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας, όπως είπαν ήδη οι συνάδελφοί μου. Είναι ένα από τα βασικά μας καθήκοντα να φροντίζουμε τον ορίζοντα 2020. Κάθε χρόνο έχουμε πολλά προβλήματα με αυτό το θέμα. Όπως γνωρίζουμε, ε, πολλά κράτη-μέλη έχουν κάνει περικοπές ε, ε, δημοσιονομικές για την εκπαίδευση και την έρευνα. Επομένως, το πρόγραμμα Ορίζον 2020 αντιμετωπίζει όλο και περισσότερα προβλήματα, όμως είναι όλο και περισσότερες οι αιτήσει κάθε χρόνο. Ξέρετε τη σημασία της βασικής έρευνας όταν τα κράτη-μέλη ε, προβαίνουν σε ε, περικοπές στον προπολογισμό τους, συνήθως πλήττει αυτό την βασική έρευνα και με απασχολεί εμένα αυτό πολύ. Όπως ξέρετε, η Ευρώπη ήθελε να είναι η πιο ανταγωνιστική, το πιο, το πιο, το πιο ανταγωνιστική περιφέρεια ε, παγκοσμίων, αλλά βλέποντα τα προβλήματα που έχουμε με το ορίζοντα 2020, ε, όπως επίσης και ε, την ιεράρχηση, τη, τη βαθμολόγηση των, των πανεπιστημίων και τη λίστα και τη λίστα της Σανγκάης δεν νομίζω ότι τα καταφέρνουμε και θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας. Τι μπορούμε να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε ότι οι ερευνητές μας έχουν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για να δουλέψουν. Θέλουμε να έχουμε ως το δυνατόν καλύτερη έρευνα στην Ευρώπη. Είναι όμως μόνο ε, το θέμα, ε, ε, θέμα χρηματοδότησης ή υπάρχουν και άλλα πράγματα που χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ την καθηγήτρια κυρία Τόλιτς. Εγώ είμαι Κροάτης, σα. Και νομίζω ότι έχω δίκιο όταν λέγω ότι πρώτη φορά έρχεται ένας τέτοιος επιστήμονας από τη χώρα μου γιατί συνήθω έρχονται πολιτικοί. Χαίρομαι λοιπόν που είναι εδώ μαζί μας κάποιος ο οποίος δείχνει ότι παρότι είμαστε μικρή χώρα με λίγα χρήματα για την εκπαίδευση και την επιστήμη σε σχέση με άλλες χώρες μπορούμε να πετύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα στην έρευνα και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι γι' αυτό. Μια μικρή ερώτηση. Σύντομη μπορεί να είναι η απάντησή σας για τις μελλοντικές σας φιλοδοξίες. Θέλετε να αγοράσατε ένα νέο μικροσκόπιο και θα ήθελα να μάθω επίσης και τι ευχές ε, έχετε για το μέλλον, τι επιθυμείτε να κάνετε στο μέλλον. Μπορώ να πω και σε ιδιωτική ε, βάση αλλά και δημοσίως ότι εμείς Λέμε μερικές φορές ότι η ομορφιά και η εξυπνάδα δεν συμβαδίζουν. Είστε η απόδειξη ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Η κυρία Σουίτσα είναι η επόμενη ομιλήτρια. You Χαίρομαι που έχουμε πάλι και εγώ μια συμπατριώτησα. Για μια ακόμη φορά σας ευχαριστούμε που οργανώσατε τη συγκεκριμένη συνάντηση. Ευχαριστώ τον κύριο European Research Council Τον ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Μποργινιόν που επέλεξε δύο εξαιρετικούς νέους επιστήμονες για να συμμεριστούν τις απόψεις σας μαζί μας. Χάρη στο Horizon 2020 τους ακούσαμε και περιμένουμε να προωθήσουν και την έρευνά τους σε επίπεδο βασικό. Όπως είπε ο συνάδελφος, δεν υπάρχουν πολλά προγράμματα από τις νέες χώρες. Εμείς έχουμε τώρα μέλη από τη νεότερη, την πιο πρόσφατη χώρα μέλος και εύχομαι κάθε επιτυχία στην κυρία Τόλιτς που είναι ανάμεσά μας εδώ και εύχομαι καλά αποτελέσματα στην έρευνά σας. Είμαι ευτυχής, είμαι υπερήφανη και συγχαίρω και εσάς, αλλά μέσω ε, ε, ημών συγχαίρω όλους όσους συμμετέχουν σε αυτά τα θέματα της έρευνας, γιατί χωρίς την έρευνα δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχει ανάπτυξη, έχει μεγάλη σημασία να επενδύει κανείς στην έρευνα, γιατί έτσι μόνο θα αντιμετωπίσει ε, τον ανταγωνισμό. Η κυρία Τόγια. Να συγχαρώ και εγώ τους δύο νέους ε, επιστήμονες και τους δύο ερευνητές. Επαναλαμβάνω το ερώτημα του κυρίου Ρόιλ. Τι μπορούμε εμείς να κάνουμε. Ευχαριστούμε για αυτήν εδώ την παρουσίαση για το 5.000 προγράμματα. Πώς μπορούμε εμείς να είμαστε πιο αποφασιστικοί. Ποιους μπορούμε να πείσουμε γιατί πολλά από αυτά τα οποία έχουμε κάνει και στα πλαίσια του Horizon μερικές φορές συναντούν πάρα πολλές δυσκολίες. Στα πλαίσια της πραγματικότητας της έρευνας υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία δεν πηγαίνουν ακόμα καλά. Τι πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο φροντίζετε εσείς το θέμα της κυκλοφορίας των ερευνητών. Γιατί πολλές φορές είστε μέσα σε έναν χώρο θα έλεγα και σε ένα θέμα πάρα πολύ συγκεκριμένο και υπερπροστατευμένο ε, τι γίνεται με την κυκλοφορία, με την επικοινωνία όταν έχετε κάνει βήματα στην έρευνα. Ευχαριστώ πολύ. Μπάνκοβιτς. Σας ευχαριστώ πρόεδρε Μπούζακ. Ευχαριστώ και την καθηγήτρια Τόλιτς και συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά για την υποτροφία σας. Έχω δύο σημεία. Πρώτον, όχι μόνο εκπροσωπείται κυρία Τόλιτς την αριστεία σε επίπεδο uh, αλλά εκπροσωπείται και την κινητικότητα των νέων, ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση Uh, Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει την κυκλοφορία των επιστημόνων, των νέων επιστημόνων. Πηγαίνει κανείς σε μια άλλη χώρα και επιστρέφει στη χώρα του για να εκμεταλλευτεί αυτά τα οποία έμαθε και το παράδειγμά σας είναι πάρα πολύ σημαντικό κυρία Τόλιτς για τους νέους βλέποντας και τις δυνατότητες για την εξήλιξη του προγράμματός σας νομίζω ότι θα συνεισφέρετε ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της έρευνας στην Κροατία. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια. Mm. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Θα ήθελα και εγώ να κάνω δύο-τρεις ερωτήσεις ε, 13 δισεκατομμύρια για θεμελιώδη έρευνα στον ορίζοντα 2020 ε, ε, από τα 17 δισεκατομμύρια για το σύνολο της έρευνας. Κατά τη γνώμη σας είναι μια καλή αναλογία. Αναλογικά δηλαδή με ενδιαφέρει, γιατί είναι πολύ λιγότερο από 20%. Άρα 70 δισεκατομμύρια ήταν το νούμερο. Ζητώ συγγνώμη. Ε, κατά τη γνώμη σας λοιπόν, ίσως να γνωρίζετε περισσότερα πράγματα για τις στατιστικές, πώς έχουν σε κάθε κράτος μέλος. Για τους νέους επιστήμονες μας, ε, όταν ε, επισκέφτεστε ερευνητικά εργαστήρια και πανεπιστήμια εντός και εκτός Ευρώπης, είμαστε αρκετά ελκυστική. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα εργαστήριά μας, το, το πνεύμα της έρευνάς μας ε, ε, στην Ευρώπη εν συγκρίση με ε, τα αντίστοιχα άλλων υπήρων πιο ελκυστική, λιγότερο ελκυστική, πώς μπορούμε αυτό να το βελτιώσουμε. Και το ερώτημα βέβαια που έθεσαν και πολλοί άλλοι συνάδελφοι πώς μπορούμε να ε, αλλάξουμε τα πράγματα, εμείς πώς μπορούμε να σας υποστηρίξουμε. Είμαστε αρκετά ελκυστικοί, γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μην χάνουμε τα ταλέντα μας, να μην φεύγουν τα ταλέντα μας, ε, ε, να μην φεύγουν σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στην Κίνα. Αυτά ήθελα να ρωτήσω. Μπορώ να σας δώσω το λόγο, κυρία καθηγητά, για να μας απαντήσετε. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να τα πω στον κύριο Όλο. Φυσικά η κατάσταση τη έρευνα σε διάφορε χώρε στην Ευρώπη διαφορετική. Υπάρχουν χώρε και η Γερμανία αποτελεί ένα καλό παράδειγμα όπου η πρόθεση τη έρευνα είναι πολύ υψηλή. Το ίδιο και στη Φιλανδία και σε άλλες χώρες, όμως είναι αλήθεια τα τελευταία χρόνια σε κάποια κράτη-μέλη η οικονομική κατάσταση οδήγησε σε περικοπές στην ε, χρηματοδότηση της έρευνας. Αλλά είδαμε σε κάποιες χώρες ότι ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο για τους ε, επιστήμονες να ε, συνεχίσουν το έργο τους καθώς οι περικοπές τους άγγιξαν κατά πολύ. Έχουμε αυτή την ιτερότητα στην Ευρώπη Υπάρχει αυτή η στήριξη από την Επιτροπή και ήταν πολύ σημαντική και η στήριξη από το Κοινοβούλιο τόσο για την ύπαρξη του ERC αλλά και για το επόμενο πρόγραμμα για το οποίο πήραμε αρκετή χρηματοδότηση. Είμαι πεπισμένος ότι θα έχουμε αυτή τη στήριξη. Όμω, η κατάσταση των ερευνητών σε διάφορες χώρε αλλάζει κατά πολύ όταν αλλάζει και η εθνική χρηματοδότηση. Από χρόνο σε χρόνο αλλάζουν τα πράγματα και αυτό πρέπει να τα παρακολουθούμε ώστε να δούμε τι θα κάνουμε. Εκλείπει η υποστήριξη στις χώρες μέλη, στα κράτη-μέλη. Αυτή η διαφοροποίηση που υπάρχει από χώρα σε χώρα συνδέεται με τις περικοπές αλλά έχει να κάνει και με το διαθέσιμα κονδύλια που υπάρχουν στα κράτη-μέλη, τα οποία είναι πολύ χαμηλά. Όσον αφορά το μέλλον, ελπίζουμε ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα. Προς το παρόν όμως, αυτή η ανισότητα που υπάρχει στα κράτη-μέλη και στη χρηματοδότηση κάνει περίπλοκη την πολύπλοκη τη ζωή των ερευνητών. και το θετική δήλωση που κάνετε για το ERC. που δεν χρειάστηκε να δώσουμε υποστήριξη στο FC είναι καλή είδηση. Δεν ισχύει μόνο αυτό για το ERC και για το Marie Curie και για κάποια άλλα προγράμματα όπως τα Widening. Αλλά πολλά πράγματα δεν έχουν αποδεσμευτεί από την χρηματοδότηση του ΕΦΣΥ. Αυτό θα είναι προβληματικό για το μέλλον και πρέπει να δούμε αν μπορούν ναι, να, επιστρεφούν έρευνα από αυτό το ταμείο στην έρευνα. Ήταν ξεκάθαρη η απόφαση για το Marie Curie ε, και άλλα ιστοτήτα αυτή δεν, δεν υπάρχει. Και το μότο μου είναι ότι εισφορά, χωρίς... Ε, ναι, το μότο μου είναι ότι αν δεν έχεις όφελος δεν συνεισφέρεις. Είναι ένα ανοιχτό ερώτημα, θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Κύριε Μούντι, σας ευχαριστώ για τη στήριξη. Θα προσπαθήσω Είμαι μαθηματικό όπω ξέρετε, ε, ασχολούμαι με γεωμετρία και ω πρόεδρο του ERC γνωρίζω... Αναγνωρίζω την ανάγκη που υπάρχει ε, και πράγματι μπορώ να σας πω ότι αυτές είναι οι συνθήκες οι οποίες θα επιτρέψουν τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη και για την ιδιωτική έρευνα. Δεν μπορεί κανείς να στραφεί μόνο στη βασική έρευνα. Δυστυχώς κάποιες χώρες αποφάσισαν το αντίθετο. Αποφάσισαν να με τον δικό τους τρόπο την έρευνα α, εκ των άνω προς τα κάτω. Κάτι το οποίο συνδέεται με ε, γρήγορη οικονομική απόσβεση. Αυτός δεν είναι ο σωστός δρόμος για να αποφύγουμε εδώ κάποιες πιθανές συγκρούσεις με συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες θα μιλήσω για τον Καναδά όπου υπήρξε η δυνατότητα ανταλλαγής επιστημόνων και οι απαντήσεις που πήρα από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας είναι ότι δεν ενδιαφέρονται γιατί ε, δεν εργάζονται με τέτοιου είδους μεθόδους. Ήταν απαγοητευτικό, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Το ίδιο ισχύει και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη φορά. Ο κύριος Μπούζεκ με ρώτησε ποια είναι η σωστή συνταγή. Ε, νομίζω ότι συμφωνούμε, νομίζω ότι το 70% θα είναι σωστό ποσοστό. 30% ε, συγγνώμη θα είναι το σωστό ποσοστό. Σε κάποιες χώρες είμαστε κοντά αλλά σε άλλες χώρες είμαστε πάρα πολύ χαμηλά. Είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι μπορεί άμεσα να υποδείξει κανείς τους ερευνητές τον τομέα στον οποίο θα αναλάβουν δράση. Να πω ότι στα πλαίσια του Horizon 2020, ακόμα και αν δει κανείς και τους άλλους πυλώνες, που δεν είναι τόσο ανοιχτοί όσο εμείς, ο τομέας της αριστείας, και αν δει κανείς τις κοινωνικές προκλήσεις Υπάρχουν πάντα δυσκολίες, αλλά υπάρχει κάποια δυνατότητα για προτάσεις εκ των κάτω προς τα πάνω. Νομίζω βέβαια ότι γενικότερα ο τομέας στα πλαίσια του οποίου κάποιος μπορεί να κάνει τις προτάσεις είναι περιορισμένος. Πάντως το Horizon 2020 δίνει δυνατότητες. Οι, οι ερευνητές ίσως να μην έχουν πλήρως συνειδητοποιήσει τις δυνατότητες ελευθερίας Τώρα κυρία Μούντι για την ερώτησή σας. Εγώ νιώθω μια κάποια απογοήτευση γιατί σαν πρόεδρος του Συμβουλίου δεν εκτίθεμαι αν θέλετε σε άλλες εξελίξεις ε, στα πλαίσια του Horizon 2020 και αυτό είναι ένα σχόλιο που έκανα στον Επίτροπο. Είναι δική του ευθύνη και όχι δική μου. Αλλά πιστεύω όμως το να υπάρχει μια σωστή δυνατότητα, τακτική δυνατότητα να συναντώμεθα είναι θετικό. Εγώ δεν θέλω να παρέμβω σε αυτά τα οποία κάνουν οι άλλοι. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα το πού βρισκόμαστε και αν υπάρχουν συνέργειες τις οποίες μπορούμε να προωθήσουμε. Είπαμε αυτό δεν είναι δική μου ευθύνη και το αναφέρω σαν κάτι το οποίο πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημασία για το σύνολο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αυτά είναι τα σχόλιά μου τώρα. Για τον κύριο Ρόιλ. Ρωτήσατε για τα επόμενα βήματα της εξελίξης. Έχουμε ε, συζητήσει πολλά από αυτά τα θέματα σε επιστημονικό επίπεδο και και διευρύνουμε τη δυνατότητα ότι ίσως θα πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο ε, σε ε, διατομιακό επίπεδο και προς αυτή την κατεύθυνση σκεφτόμαστε ε, ε, ότι δεν είναι παρκές να καλύπτουμε μονάχα το κομμάτι του engineering. Θα πρέπει να σκεφτούμε κάτι παραπάνω και ενδεχομένω τα επόμενα χρόνια να υπάρξουν νέα πάνελ προς την κατεύθυνση του engineering για να υπάρχει μεγαλύτερη ομογένεια. Αυτό θα βελτιώσει την ποιότητα του έργου όταν θα μπορέσουμε να καλύψουμε τους διαφορετικούς ε, τομείς με ρωτήσετε και για το widening που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Μόλις ανέλαβα την Προεδρία κάναμε, δημιουργήσαμε μια ομάδα εργασίας. Ήταν μια πρόταση που εγκριθήκε από πολλά μέλη από το Επιστημονικό Συμβούλιο και αυτά που έχουν γίνει μέχρι στιγμής και πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Ε, τρία σημεία ένα ερωτηματολόγιο που το στείλαμε σε ερευνητέ και συγκεκριμένα σε ερευνητέ χωρών που δεν έχουν πολλέ υποτροφίε. που παίρνουν υποτροφίε εκτό τη χώρα του και να μα εξηγήσουν ε, ικανοποιημένοι με την κατάσταση, τι μπορούν να μα προτείνουν κτλ. Και επίση να δώσουμε την ευκαιρία να δώσουμε την ευκαιρία να αναφέρουν τι ήταν καθοριστικό για τη μετακίνησή τους και φυσικά το ερώτημα για τη διαθεσιμότητα χρημάτων είναι πολύ σημαντικό, όμω αυτό που είδαμε ήταν ότι υπήρξαν και άλλα προβλήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την τεχνική, τεχνολογική, τεχνική υποστήριξη που έχουν ειδικά από διοικητική πλευρά. Επίσης, ε, η ακαμψία του συστήματος που δεν επιτρέπει γρήγορες αντιδράσεις είναι πολύ επισημαντικό για τους ερευνητές. Θέλουν να μπορούν να προσελκύουν στις ομάδες τους ερευνητές ε, Ερευνητέ ε, εξωτερικούς και σε κάποιες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση το να το κάνουν αυτό είναι πολύπλοκο. Τόσο πολύπλοκο που όταν είσαι στη θέση να το κάνεις, το άτομο που θέλεις να προσλάβεις έχει ήδη αποχωρήσει γιατί έπρεπε να περιμένει πολύ καιρό. Υπάρχουν εμπόδια, κάποια είναι οικονομικά σίγουρα και φυσικά όταν μια χώρα δεν επενδύει πολύ στην έρευνα τότε αυτό αποτελεί μεγάλο μειονέκτημα για την έρευνα. Ένα άλλο κομμάτι έχει να κάνει ε, με τον ε, αριθμό ε, με, τον, με την απασχόληση των ερευνητών και τους μισθούς τους γιατί πολλοί αναγκάζονται να εργάζονται και σε άλλες δουλειές και δεν έχουν τόση ενέργεια για να αφαιρώσουν στην έρευνα. Επίσης γίνεται προσπάθεια από κάποιες χώρες που είναι να δοθεί η δυνατότητα σε ερευνητέ. Υπάρχει μια πρωτοβουλία σχετική από την Πολωνία και την Ουγγαρία, αλλά ελπίζουμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλε χώρε. Να έχουν λοιπόν τη δυνατότητα ερευνητέ, συγκεκριμένα νέοι ερευνητέ, να επισκέφτονται ομάδε του ERC για λίγου μήνε, ώστε να δουν πώ είναι οργανωμένε και να προετοιμαστούν για μια μελλοντική αίτηση. Τη ιδέα μια σύντομη εκπαίδευση ώστε να δούμε πώ γίνονται τα πράγματα θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα. Και το τελευταίο σημείο που θέλω να αναφέρω είναι κάτι για το οποίο θα δώσει οικονομική στήριξη στο ARC άμεσα. Είναι ένα πρόγραμμα που θα υποβληθεί από τις εθνικές αρχές επαφής για την οργάνωση και τη βοήθεια στο επίπεδο αλληλεγγύης ώστε να βοηθηθούν οι ερευνητές στη συνεργασία και ειδικά ε, ερευνητές από χώρε που δεν έχουν τόσο μεγάλη επιτυχία για να μπορέσουν να προετοιμάσουν τις αιτήσει τους. Υποβλήθηκε λοιπόν ένα πρόγραμμα από, από τις Εθνικές Αρχές Επαφής και για το 2016 έχουμε ε, δεσμεύσει συγκεκριμένο αριθμό, συγκεκριμένα κονδύλια για αυτό το πρόγραμμα. Το, ε, παίρνουμε πολύ σοβαρά αυτό το θέμα. Δεν ε, περιμένουμε άμεσα αποτελέσματα, θα χρειαστεί λίγος χρόνος. Όμως είναι κάτι που θέλουμε να ε, βελτιώσουμε. Ο ρόλος της κατάταξης ήταν μια ερώτηση που μου τέθηκε και είπα ότι δεν ήταν το μόνο πρόβλημα τα χρήματα, αλλά ήταν και το θέμα της ευελιξίας η οποία είναι απαραίτητη και ως μαθηματικός αισθάνομαι ότι ο ρόλος του ranking της κατάταξης είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε πολύ, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Υπάρχουν πολλές υπηρεσίε που δεν ε, ε, βασίζουν ε, την κρίση τους μόνο στο ranking αλλά και στα bibliometrics στα μαθηματικά, στον κλάδο μου τα bibliometrics δεν είναι καθόλου χρήσιμα. Όμω έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ αυτό ο κλάδο που έχει γίνει σχεδόν δικτατορία. ω πρόεδρο του ERC και αυτοί με ακούνε, ενημερώνουν τα μέλη των πάνελ και τα επαναλαμβάνω με κάθε ευκαιρία γιατί θέλω τα μέλη του πάνελ να δουν ε, τα αποτελέσματα και την ποιότητα των ερευνών και να μην αποφασίζουν ε, ε, ότι κάποιος είναι καλύτερος από τον άλλον εξαιτίας αυτών των ε, rankings. Είναι μια παγκόσμια προσπάθεια που πρέπει να καταβάλουμε. Είναι καλό φυσικά να υπάρχει κρίση, να κρίνεται το έργο μας, αλλά η μείωση αυτών των κριτηρίων ε, θα είναι αρνητική για δραστηριότητε όπω ε, και για τα πανεπιστήμια που πρέπει να είναι πολύ ενεργά στην έρευνα, πρέπει να είναι στην κορυφή τη έρευνα. Να είναι αποδοτική όμω και στη διδασκαλία. Πώ θα διαχωρίσουμε αυτά τα δύο, Είναι ένα. Ε... Innovation. So that's the third dimension. How can you reduce this to just one number? It doesn't make sense. So you have to um, approach these questions uh, with a very uh, broad approach. And to finish with the question of uh, Mrs. Toya, je vais revenir Français, si vous me permettez. Euh, donc, euh, Έχω την αίσθηση ότι τα πολύ σημαντικά για το Ταμείο μας, για το Ινστιτούτο μα, αν θέλετε, το Συμβούλιο μας, είναι να συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση, να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στα πλέον φιλόδοξα σχέδια, στα οποία αναλαμβάνουμε κινδύνους αλλά περιμένουμε να υπάρξει απόδοση, και κάνοντας την επιλογή αυτή πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τον αριθμό των δημοσιεύσεων γιατί αν τα σχέδια αυτά είναι νέα πρόσφατα θα απαιτήσει αρκετό χρόνο κάτι τέτοιο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν σε τέτοιου είδους υπολογισμούς με τον αριθμό των δημοσιεύσεων μόνο. Πάντως το Horizon 2020 λέγει ότι όλες οι χρηματοδοτήσεις οι ευρωπαϊκές θα πρέπει να είναι ελεύθερης πρόσβασης. Αυτό έχει κάποιες συνέπειες. Νομίζω οι επιστήμες μπορεί να είναι εύκολες ή δύσκολες, οι κοινωνικές επιστήμες όπου οι δημοσιεύσεις είναι βιβλία και τα βιβλία χρειάζονται χρόνο και το σχήμα χρηματοδότησης κάνει όταν ολοκληρωθεί το Συμβούλιο να μην υπάρχουν χρήματα. Οπότε πώς θα βοηθήσουμε για τη δημοσίευση των βιβλίων ε, τους ερευνητές οι οποίοι έχουν τύχει στήριξης για να προετοιμάσουν τα βιβλία αυτά και θα πρέπει να τα θέσουν σε ελεύθερη πρόσβαση τη στιγμή κατά την οποία δεν έχουν τα χρήματα να το κάνουν. Είναι ένα τεχνικό θέμα το οποίο χρήζει επίλυσης γιατί πράγματι είναι εντελώς παράλογο με, με ακατάλληλη χρηματοδότηση να πιέζουμε τους ερευνητές της κοινωνικές επιστήμες να δημοσιεύουν με μικρά άρθρα και όχι με ένα ολοκληρωμένο κάθε φορά πόνημα. Ευχαριστώ τον καθηγητή Μπουργκινιόν για όλες τις παρατηρήσεις του και τις εξηγήσει του. Έχετε το λόγο, κυρία Τόλιτς. Ε, φυσικά ανησυχώ για τις περικοπές και οι συνάδελφοι ανησυχούν για τις περικοπές. Εγώ για τα επόμενα χρόνια λόγω του Συμβουλίου και κάποιων μικρότερων επιδοτήσεων και υποτροφιών καλύπτομαι τι θα γίνει μετά τα επόμενα χρόνια πέντε δεν ξέρω. Ελπίζω να υπάρξουν πιστώσεις για τους νέους ερευνητές. Το όνειρό μου επιστημονικά είναι να κατανοήσω το πώς διαιρούνται τα κύτταρα και να δημιουργήσουμε ένα κέντρο για το είδος της φυσικής το οποίο έχει σχέση με την βιοφυσική και να αναγνωριστούμε σε παγκόσμιο επίπεδο έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι ότι αυτή η διεπιστημονική έρευνα σε επίπεδο διέρεσης κιτάρων διεξάγεται με επιτυχία στο Ζάγκρεμπ. Το Ινστιτούτο Μπόσκοβιτς έχει επίσης από από άλλα προγράμματα ε, βοηθηθεί οικονομικά και έχει δημιουργήσει θέσεις έρευνας και έχει προσκαλέσει και άλλους επιστήμονες ε, της δικιάς μου γενιάς στην Κροατία πίσω. Υπάρχει λοιπόν το απαιτούμενος αριθμός για την διεξαγωγή της έρευνας και το μέλλον εδώ ε, είναι αρκετά ρόδινο. Αυτό το πετυχαίνω γιατί έκανα την καριέρα μου μέχρι τώρα στην Γερμανία, είχα εξαιρετικές συνθήκες, ευκαιρίες, συναδέλφους στο Max Planck και νομίζω ότι οι άνθρωποι της γενιάς μου που έχουν περάσει τον περισσότερο χρόνο τους στο Ζάγκρεμπ είχαν δυσκολίες μπροστά τους, δεν μπόρεσαν να, να δουλέψουν σωστά και δεν είχαν και το ε, βιογραφικό που θα τους επέτρεπε να πάρουν την υποτροφία του Ευρωπαϊκού αυτού Ταμείου. Πρέπει να υπάρξει βοήθεια για πιλωτικά προγράμματα και την βελτίωση του βιογραφικού των επιστημόνων. σχετικά με το πόσο ελκυστική είναι η Ευρώπη είναι να υπάρξουν καταρχάς περισσότερες μόνιμες θέσεις, πάρα πολλά ευρωπαϊκά όργανα δεν έχουν τέτοιου είδους δυνατότητες σταδιοδρομίας. Είναι καλό για τους οικοσάριδες να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά σε διάφορες χώρες, αλλά όταν φτάσουν τα 30 και μετά οι περισσότεροι θέλουν κάπως να σταματήσουν να μετακινούνται. Θα ήταν ελκυστικό λοιπόν και για τους εκτός Ευρώπης αν τα Ινστιτούτα και τα Πανεπιστήμια μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερες μόνιμες ή σχετικά μόνιμες θέσεις. Συν βέβαια τις επιδοτήσεις για έρευνα. Και για τις γυναίκες στην επιστήμη το Συμβούλιο δίνει την δυνατότητα υπέρβαση αν θέλετε μετά από χρόνια στην συγγραφή του διδακτορικού για λόγους μητρότητας. Είναι πολύ ενδιαφέρον και καλύπτει τις ανάγκες γυναικών. Καλό θα ήταν να υπάρχουν ειδικέ διευκολύνσεις και για γυναίκες με παιδιά για να μπορέσει ο κόσμος να εργαστεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Πούνια. για την ερώτηση της κυρίας Τόγια που είπε τι μπορούμε να διορθώσουμε. Προσωπικά εγώ υποχρεώθηκα να μεταφέρω την επιδότηση αυτή από το ένα πανεπιστήμιο στο άλλο. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να βελτιωθεί η μεταφερσιμότητα θα έλεγε κανείς της, ε, της συγκεκριμένης χρηματοδότησης. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Ε, τα βασικότερα θέματα τα έθεσε ο κύριος Μπουργκινιόν. Ε, χρειάζεται ένας κατάλληλος προϋπολογισμός για να προεθηθούν τα προγράμματα. Υπάρχουν τεράστιες ανάγκες, ζούμε εθνικές συνθήκες δραματικού τύπου θα έλεγα και ακόμα και όταν υπάρχουν χρήματα είναι δύσκολο να κατανεμηθούν με σωστό τρόπο. Το θέμα είναι όχι μόνο οι πτυχιούχοι βέβαια, αλλά και αυτοί οι οποίοι κρίνουν τις προτάσεις. Εμείς παίρνουμε πάρα πολλά σχόλια από σχολιαστές επιστημονικών δημοσιεύσεων. Πολλές φορές υπάρχουν διαφορές στις απόψεις αφές, αλλά νομίζω ότι και οι στατιστικές δείχνουν ότι πάντα υπάρχει στο τέλος συμφωνία σε σχέση με τον χαρακτηρισμό των προτάσεων. Έτσι διασφαλίζεται μια σωστή χρηματοδότηση η οποία σε μια θα έλεγα περίοδο κρίσης, δεν θέλω να μιλάω πάντα για κρίση γιατί η κρίση έχει και θετικά τελικά στοιχεία αλλά έχει σημασία αυτού του είδους οι χρηματοδοτήσεις να συνεχιστούν. Τώρα για την διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας θα συμφωνήσω με αυτά τα οποία έλεγε ο πρόεδρος ότι σήμερα η βιβλιομετρία έχει καταστεί μια δικτατορία, ο αριθμός των δημοσιεύσεων δηλαδή. Ε, Βασικό ε, βασικός στόχος των επιστημόνων είναι να δημοσιεύει ε, άρθρα. Νομίζω ότι εγώ πάρα πολύ συχνά πηγαίνω σε ε, διάφορες συναντήσεις και σε αίθουσες μεγάλες για να παρουσιάζω τις εργασίες ε, της ομάδας μου και τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών. Τώρα για τις συνεργασίες, ε, νομίζω εν μέρη έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις. Να πω ότι όταν κάποιος παίρνει ένα μια τέτοια επιδότηση, η οποία είναι ad personam καταρχάς, νομίζω ότι αυτό ε, καλύπτει ένα ευρύτερο πεδίο έρευνας γιατί εμείς στην προσπάθειά μας όπως είπα συνεργαζόμεθα ε, με ε, μια μεγάλη ομάδα και επιχειρήσεων στην Ευρώπη που έχουν ηγετική θέση αλλά και άλλους επιστήμονες. για τη βασική έρευνα. Η βασική έρευνα είναι πολύτιμη, είναι θεμελιώδης, δεν υπάρχει πραγματικά... Μπορεί να πει κανείς ότι η βασική έρευνα είναι η προϋπόθεση για οτιδήποτε άλλο. Και χθες που ήρθα στις Βρυξέλλες συνάντησα μια βιομηχανία η οποία ενδιαφέρεται για έρευνες με τις οποίες ασχολούμαι, βασικές έρευνες οι οποίες αύριο μπορεί να βρούνε εφαρμογή. Σας ευχαριστώ κύριε Μπουργκινιόν, ευχαριστώ και τους δύο επιστήμονες για την επίσκεψή σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για μας να σας συναντήσουμε και να συζητήσουμε. Θα θέλαμε λοιπόν εμείς με βάση αυτά τα οποία είπατε στην έρευνα και στην καινοτομία και στη βασική έρευνα η οποία είναι απαραίτητη για κάθε τύπου καινοτομία για τα επόμενα 5-10 χρόνια και γι' αυτό ακριβώς η επίσκεψή σας ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για όλους μας. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά. Η επόμενη συνάντησή μας τελειώσαμε βέβαια. 23 η Ιουνίου από τις 3 μέχρι τις 6.30 το απόγευμα.